Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω σε αυτό το εργαστήριο. Καταρχάς να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτικής ΕΝΤΗ και το Τμήμα Προϋπολογισμού για την πολύ καλή διοργάνωση. Καλωσορίζω επίσης και τους εμπειρογνωμονές μας, οι οποίοι έχουν έρθει για να μας ε, παρουσιάσουν το θέμα αυτό. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων είναι για την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι τα έσοδα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων αποκρύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και από τον Προπολογισμό των ε, κρατών μελών. Είναι διαφυγόντα λοιπόν κέρδη και οι πληροφορίε μας λένε ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων έχει αυξηθεί σημαντικά κάτι που αφορά επίσης ε, και την, ε, τον τομέα της υγείας. Παρότι έχει ε, φανεί ότι έχουν μειωθεί η κατανάλωση τσιγάρων, ωστόσο το, οι πληροφορίε μας λένε ότι το 1 στα 5 τσιγάρα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελαθρέο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι χάνει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδος το ποσό αυτό για την Γερμανία για το έτος 2012 ανέρχεται στα 870 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ψηλό ποσό και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θεώρησε καλό να ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα αυτό. Πρωτού δώσω το λόγο στον ε, Μπαρτ Στές, τον ε, εισηγητή και αντιπροθέτη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θα ήθελα καταρχάς ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού να καλωσορίσω τους ομιλητές. Η πρώτη ομιλήτρια θα είναι καθηγήτρια Άννα Γκίλμορ από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα μας παρουσιάσει μια επισκόπηση της κατάστασης από επιστημονικής πλευράς. Ο δεύτερος ομιλητής δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει, ο Άμιρ Λατίφ. Έπειτα, ο τρίτος ομιλητής θα είναι ο Κύριο Σεπιού από την Ευρωπόλ, καλώς ορίσατε. Η Ευρωπόλ καθώς και ο Όλαφ δραστηριοποιούνται ενεργά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και βρίσκονται στη μέση της αίθουσα και μας έχουν φέρει πληροφορίες για στατιστικά στοιχεία σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λέσεκ Παρτολομιέτσικ από τη Βαρσοβία της Πολωνίας, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Καλώς ήλθατε. Επίσης τον κύριο Λουκ Γιώσενς, την Χάνα Ρος και τον κύριο Στοκ Λόσα που θα μιλήσουν αργότερα και τέλος την συνάδελφο κυρία Ίνκε Κρέσλε. Θεωρήσαμε ότι λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μεγάλη παρουσία συναδέλφων, όμως όσοι είστε εδώ σίγουρα έχετε δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα, το οποίο συνδέεται και με την ψηφοφορία για την οδηγία για τον καπνό, η οποία θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται μόνο εδώ και λίγο καιρό με το θέμα αυτό, με το λαθρεμπόριο τσιγάρων, αντίθετα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Πιστεύουμε πως έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, ασχολούμαστε εδώ και πολύ καιρό και γι' αυτό και ευχαριστούμε και όλους μας τους συνεργάτες. Λοιπόν, σας καλωσορίζω άλλη μία φορά. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση είναι ανοιχτή, μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Έχουμε διερμηνία σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάρτ Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε όλοι, καλώς όρισαν όλοι οι προσκεκλημένοι, οι εμπειρογνώμονες. Και βεβαίως επανέρχομαι σε αυτό που μόλις είπε ο Πρόεδρος. Αυτή η ακρόαση ουσιαστικά επιτρέπει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού να συνεχίσει μια μακρόχρονη παράδοση. Το θέμα της καταπολέμησης της απάτης είναι κάτι που μας απασχολεί. Ήδη από τη δεκαετία του 90 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ειδική διερευνητική επιτροπή για να ασχοληθεί με το θέμα ακριβώς αυτό της ε, καταπολέμησης της απάτης και μάλιστα τότε είχαμε πάρει μεταξύ άλλων παραδειγμάτων και το θέμα του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και πριν ιδρυθεί Όλαφ, ο προηγούμενος οργανισμός, ο προκάτοχος του Όλαφ, ο Κλαφ είχε επίσης ασχοληθεί με το θέμα αυτό στον προηγούμενο αιώνα, στο τέλος του 20ου αιώνα και πολλά είχε κάνει τότε ο οργανισμός αυτός, ο προκάτοχος ε, του Όλαφ για να διερευνήσει το θέμα αυτό και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που είχαν εργαστεί ε, στα πλαίσια αυτού του οργανισμού και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτοί που ξεκίνησαν αυτές τις έρευνες. Επίσης θα ήθελα εδώ να αναφέρω και την καπνοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τσιγάρων που πραγματικά σε συνεργασία μαζί μας μας δίνουν πολύ σημαντικά στοιχεία, κάτι που μας επέτρεψε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ να επανέλθουν στα κρατη να επανέλθουν στους προϋπολογισμούς του και περίπου το 9,7% από αυτό το ποσό έχει χρηματοδοτήσει μία σειρά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Επίσης, προγράμματα για την καλύτερη συνεργασία των τελωνιακών αρχών. Τι άλλο όμως κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά τα κονδύλια. Έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες χώρες, όπως τη δική μου, τα χρήματα αυτά δεν ε, διοχετεύονται στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας που έχει σχέση με το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Είναι απαραίτητο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε αυτήν την καταπολέμηση, διότι η απάτη αυτή, το λαθρεμπόριο αυτό, ουσιαστικά εδώ συνδέεται με άλλου είδους εγκληματικότητα. Ο Αμίρ Λατίφ δημοσιογράφος από το Πακιστάν έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο με το θέμα αυτό και πραγματικά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η βελγική πρεσβεία παραδείγματος χάρη στο Ισλαμαμπάν δεν συνεργάστηκε και δεν μπόρεσε ο άνθρωπος αυτός να είναι σήμερα εδώ. Ευτυχώς έχουμε την ομιλία του, έχουμε την παρέμβαση που θα ήθελε να κάνει και μπορείτε να την διαβάσετε. Είναι στη διάθεσή σας εδώ στην αίθουσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θεωρεί ότι το διαφυγόν κέρδος φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι ένα σημαντικό ποσό και κάθε χρόνο οι κατασχέσεις φτάνουν τα 6 δισεκατομμύρια τσιγάρα. Κάθε χρόνο και 10 εκατομμύρια ευρώ, 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το διαφυγόν κέρδος. Είναι πολύ κρίμα που τα κράτη-μέλη δεν κάνουν περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Και όταν κανείς κάνει την ερώτηση αυτή στο Συμβούλιο των Υπουργών, η απάντηση είναι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και να ξανακάνουμε ερώτηση στην ε, επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. Το πρόγραμμα Ηρακλής, μια σειρά μάλλον προγραμμάτων πολύ σημαντική, με σκοπό τον συντονισμό των μέτρων που έχουν σαν σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στήριξη. Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών, καλύτερη κατάρτιση των τελωνιακών διότι δέκα χρόνια μετά την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων ε, στον τομέα των τσιγάρων όπως της Φίλιπ Μόρις, βλέπουμε ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για να είμαστε αποτελεσματικοί. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα, διαπιστώνουμε ότι οι απόπειρες να περιοριστεί η προσφορά στη μαύρη αγορά τσιγάρων δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές. Και οι επιχειρήσεις, οι καπνοβιομηχανίες, ουσιαστικά εδώ προτιμούν να πληρώσουν ένα πρόστιμο, αλλά διαπιστώνουμε ότι τα πρόστιμα αυτά, οι κατασχέσεις αυτές είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό δείχνει ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων συνεχίζει να ανθίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε στην σημερινή μας ακρόαση πώς ο τομέας μπορεί να βρει τρόπο να αντιδράσει και πώς πολλές φορές τα τσιγάρα τα οποία είναι προϊόν κατάσχεσης δεν είναι καθόλου παράνομα τσιγάρα, είναι κανονικά προϊόντα, κανονικά τσιγάρα, τα οποία απλώς έχουν διοχετευθεί μέσω των παράνομων δικτύων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό καταρχήν να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα τσιγάρα που πολλούνται μέσω των ε, λαθρέων δικτύων, των παράνομων δικτύων, είναι πραγματικά απομιμήσεις τσιγάρων, παράνομα τσιγάρα, ω προ την κατασκευή του. Πολλέ φορέ ζητήσαμε λοιπόν από τον Όλαφ να κάνει αυτήν τη διάκριση, αν πρόκειται για αφεντικά τσιγάρα ή όχι. Και αυτό πρέπει να σα πω δεν έχει ποτέ γίνει. Η έκθεση του Ιαν Βόλτεν ακριβώς αυτό διαπιστώνει και ο Επίτροπος Σέμετα απάντησε στην ερώτησή μου λέγοντας ότι το Scottish Ocean Institute έχει ξεκινήσει μια έρευνα, πρόκειται για μια σκοτσέζικη οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ηρακλής. Στον ιστότοπό τους εγώ δεν διαπιστώνω καμία, απολύτως καμία αναφορά στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος που να αφορά τον καπνό ή τα τσιγάρα και τις παράνομες δραστηριότητες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Όλαφ έχει μειώσει, αν θέλετε, τις προσπάθειες του για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Έχει μειωθεί η εμβέλεια αυτών των ε, ερευνών, αυτών των μελετών και την ίδια ώρα βλέπουμε να συνεχίζουν οι παράνομες δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές άλλες εξηγήσει για να δικαιολογήσει κανείς ε, αυτήν την μείωση όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα του Όλαφ. Οι αποστολές παράνομων τσιγάρων σήμερα έχουν αλλάξει μορφή. Διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες αποστολές προμήθειες παράνομων τσιγάρων γίνεται με πολύ μικρά πολύ μικρές ποσότητες, που δεν ξεπερνούν δηλαδή τις 50.000 τσιγάρα. Πρόκειται ουσιαστικά για πολλές επαναλαμβανόμενες μικρές αποστολές. Και πάνω από 100.000 τσιγάρα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Αυτό ίσως δικαιολογεί το πώς έχει αλλάξει αυτή η παράνομη διάθεση τσιγάρων με τον πολλαπλασιασμό των αποστολών μικρότερων ποσοτήτων, έτσι ώστε να βρίσκονται κάτω από το όριο επιβολής των προστήμων. Με τον Λουκ Γιός, εμπειρογνώμονα από το Βέλγιο, προετοιμάσαμε μία μελέτη και όσοι διάβασαν την έκθεσή του θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι ουσιαστικά η παράνομη διάσταση τσιγάνων στην Ευρώπη συνεχίζεται ακάθαρτα, ότι οι πηγές ε, είναι η Ουκρανία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε κερδίσει μία μάχη. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες και να κατανοήσουμε καλύτερα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προοδεύσουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για να αποφύγουμε αυτές τις πολύ αρνητικές συνέπειες. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα διαφυγόν κέρδος της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα ποσά καλά θα κάνουμε να τα επαναφέρουμε στους προϋπολογισμούς. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκίλμορ όμως. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. I just want to talk about two things today. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα σήμερα στα 15 λεπτά που μου έχετε δώσει. Καταρχάς, ε, έχουμε όλο ένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι καπνοβιομηχανίες ε, συμμετέχουν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και στην παράνομη διακίνηση των προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια κυκλοφορούν παρανόμως στην αγορά. Και να σας αναφέρω και τις ανησυχίες που υπάρχουν ε, για τη στοιχεία υπάρχουν αρκετές ανησυχίες για τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν αναφερόμαστε στην κάποια βιομηχανία, αναφερόμαστε στις τέσσερις βασικές ε, ε, επιχειρήσεις, τη Philip Morris, τη Japan Tobacco, και τις άλλες δύο μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι όλο το λαθρεμπόριο τσιγαρών στην Ευρώπη οφείλεται σε αυτές τις τέσσερις επιχειρήσεις, αλλά ε, μεγάλο ποσοστό οφείλεται ε, σε αυτές και αυτό το παραβλέπουμε συνεχώς. Να σας δώσω λίγο το ιστορικό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ιστορικά για την συμμετοχή των καπνοβιομηχανιών στο λαθρεμπόριο τσιγάρων σε παγκόσμια κλίμακα. Πολλά από τα στοιχεία προέρχονται από τα ίδια τους τα έγγραφα. Έκανα μεγάλη έρευνα ε, στην τεκμηρίαση αυτή τα τελευταία 13 χρόνια και πρέπει να σας πω ότι όποια χώρα έχω εξετάσει έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν καπνοβιομηχανίες που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Επίσης, ε, το λαθρεμπόριο τσιγάρων ήταν βασικός πυρήνας ε, των εργασιών τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφηκε στο δικαστήριο και κατέληξε σε συμφωνία στη Νέα Υόρκη. Η υπόθεση διαδικάστηκε στη Νέα Υόρκη και μετά από εκεί και πέρα αρχίσαμε να βλέπουμε μια αλλαγή ε, στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Έχουμε μια πιο ανάμεικτη εικόνα, έχουμε και απομιμήσεις και τα λεγόμενα illicit whites. Είναι ε, τσιγάρα τα οποία παράγονται νόμιμα αλλά διακινούνται παράνομα στην αγορά. Υπάρχει μία αλλαγή η οποία όμως παρουσιάζεται περισσότερη από ό,τι είναι για διάφορους λόγους. Καταρχάς ε, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει παρουσία παράνομων τσιγάρων. Αυτό το έχουμε και από τα στοιχεία της Φιλιπ Μόρις ήδη. Υπάρχουν διεθνείς καπνοβιομηχανίες οι οποίες εμπλέκονται στην παράνομη διακήρυξη τσιγάρων και υπάρχουν και ενδείξεις ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την αλυσίδα εφοδιασμού και πολλές φορές διαραίουν τσιγάρα στα παράνομα κυκλώνωματα. Ο λόγος για τον οποίο τις απομιμήσεις τσιγάρων είναι ε, διότι τα δεδομένα δεν είναι αξιόπιστα και ότι τα κατασκευμένα τσιγάρα είναι πολύ περισσότερα από όσα στην πραγματικότητα φαίνονται από τα στοιχεία που έχουμε. Να σας δώσω εδώ τις αποδείξεις που έχω. Εδώ έχουμε ε, αποδείξεις ότι υπάρχει διακίνηση τσιγάρων τουλάχιστον μέχρι το 2010. Από ερευνητική δημοσιογραφία που έγινε το 2011 διαπιστώθηκε ότι ε, υπήρχε πολύ μεγάλη ανάμειξη και αν οι δικηγόροι της Japan Tobacco δεν είχαν σταματήσει την έρευνα θα είχαμε ακόμα περισσότερα στοιχεία. Υπήρχε λοιπόν εμπλοκή σε παράνομη πορεία τσιγάρων και εντός της Japan Tobacco και φαίνεται ότι δεν έκανε τίποτα η συγκεκριμένη καπνοβιομηχανία όταν τους παρουσιάστηκαν αυτές οι αποδείξεις. Απλώς ε, ε, σταμάτησαν τις έρευνες, ε, τους ε, χάκαραν τους υπολογιστές και τελικώς κατάφεραν να σταματήσουν τελείως ε, ε, διότι απολύθηκαν οι ερευνητές αυτοί. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε, η Όλαφ συγγνώμη, διαπίστωσε ότι υπήρχε διακίνηση τσιγάρων στην Συρία παρά τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Προσφάτως δημοσιεύθηκε και ένα έγγραφο για τη Βουλγαρία και υπάρχουν αρκετές πηγές που καταδεικνύουν ότι υπάρχει συνενοχή στην ε, λαθρεμπόριο τσιγάρων ε, μεταξύ του 2000 και του 2010, μετά λοιπόν τη σύναψη των συμφωνιών με τις καπνοβιομηχανίες. Προσφάτως, και θα σας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια ο συνάδελφος, έχει ε, καταστεί σαφές ότι μία από τις ε, μάρκες που διακινούνται περισσότερο είναι η λεγόμενη μάρκα Classic, που είναι ε, θεωρείται ότι είναι η λύση του Άιτ και τελικώ παράγεται από μια καπνοβιομηχανία στην Ουκρανία. Το 2009 αυτό ήταν περίπου το 7% της παράνομης ε, διακίνησης τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα της ε, υπερπαραγωγής. Ε, και πάλι από ερευνητική δημοσιογραφία διαπιστώσαμε ότι το 2008 οι καπνοβιομηχανίες αυτές παράγουν 30 ε, δισεκατομμύρια τσιγάρα περισσότερα από όσα μπορούν να καταναλώσουν οι Ουκρανοί και αυτά στη συνέχεια δεκινούνται στην παράνομη αγορά ε, της Ευρώπης. Συλλογικά όλες αυτές οι ενδείξεις ε, της υπερπαραγωγής στην Ουκρανία, της παραγωγής των παράνομων λευκών στην Ουκρανία, τη συμμετοχή στο λαθρεμπόριο τσιγάρων στη Ρωσία και τα στοιχεία τα οποία έχουμε έδειξαν ότι η Ρωσία και η Μέση Ανατολή ε, είναι ε, μπλεγμένες ε, στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Γι' αυτό και έχουμε και το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο τσιγάρων στα ανατολικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, Υπάρχει και η έκθεση Project Star της Φίλιπ Μόρις, Μετά από τη συμφωνία την οποία σύναψε η Φίλιπ Μόρις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την αγωγή η οποία κατατέθη στη Νέα Υόρκη το 2007, ε, η Φίλιπ Μόρις προσέλαβε μια λογιστική επιχείρηση για να κάνει μια μελέτη για το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να διαπιστώσουμε το βαθμό της ανεξαρτησίας αυτής της έκθεσης. Η Φίλιπ Μόρις λέει ότι το Project Star διεξάγεται από την KPMG για την Φίλιπ Μόρις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Ε, και φαίνεται όμω ο Λεώνα και περισσότερο ότι δεν ισχύει αυτό στην πραγματικότητα και ότι η έκθεση είναι ε, στην πραγματικότητα υπό τον έλεγχο τη Φίλιπ Μόρι. και θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαρκή διαφάνεια για αυτό το θέμα. Τι κάνει τώρα η έκθεση. Παίρνει μία σειρά από δεδομένα και τα ε, ε συμπεριλαμβάνει για να δια, ε, δημιουργήσει ένα μοντέλο. Έχουμε κάποια πρόσφατα στοιχεία από την έκθεση αυτή, η οποία έχει δημοσιευθεί, έχω φέρει και κάποια αντίγραφα εδώ και νομίζω ότι και το ίδιο το μοντέλο είναι καλή ιδέα και θα μπορούσε να μας δώσει χρήσιμα στοιχεία, αλλά ανησυχούμε διότι τα στοιχεία τα οποία έχουν εισαχθεί στο μοντέλο μπορεί να μην είναι ακριβή. Θα σας πω λίγα περισσότερα στη συνέχεια. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαπιστώσεις για την ε, ε, υπερπαραγωγή τσιγάρων. Η Φίλιπ Μόρις ε, δεν μπορεί να μας δώσει για παράδειγμα στοιχεία για τη διανομή για τα ελληνικά νησιά παρά το γεγονό ότι ξέρουμε ότι τα ελληνικά νησιά είναι ένας από τους χώρους στου οποίου γίνεται παράνομη διακίνηση. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να μας δώσει αξιόπιστα στοιχεία για το τι γίνεται για τη διανομή τσιγάρων εκεί. Επίσης, το μοντέλο εκτιμά ότι το 1 τέταρτο των λαθρέων τσιγάρων στην αγορά του 2010 ήταν από τι μάρκε που διαθέτει η Φιλιπ Μόρι και ε, έχουμε 5% παραποιημένα τσιγάρα της μάρκας ε, των Φιλιπ Μόρι τσιγάρων. Να σας δώσω εδώ το διάγραμμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ έχουμε τα στοιχεία του 2010. Τα στοιχεία και το 2011 είναι αντίστοιχα, δεν υπάρχουν βέβαια στην έκθεση που έχουμε. Ε, το 24% περίπου λοιπόν το 1 τέταρτο των λαθρέων τσιγάρων στην Ευρώπη είναι μάρκες της Φίλιπ Μόρις, σε σύγκριση με 5% μόνο παραποιημένα τσιγάρα. Αν δούμε τα στοιχεία του 2006, τα στοιχεία είναι 40% από τις μάρκες της Φίλιπ Μόρις και 7%. Η αναλογία είναι γύρω στο 5%. Είναι 5,7, 5,5, 5,2 στα τελευταία στοιχεία, τα πιο πρόσφατα που έχουμε. Η αναλογία λοιπόν της παραγωγής ε, της Φίλιπ Μόρις έχει ε, ε, μειωθεί και έχουμε φτάσει περίπου στο 1 τέταρτο των ε, λαθρέων τσιγάρων που είναι περίπου αυτή η παραγωγή που έχουμε στις μάρκες της Φίλιπ Μόρις. Τα κατασχεμένα όμως δεδομένα που έχουμε μας δίνουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Το στοιχείο εδώ είναι 89% στις κατασχέσεις, ότι είναι τσιγάρα της Φίλιπ Morris από μιμήσεις και μόνο 11% είναι αυθεντικά τσιγάρα της Φίλιπ Morris. Εδώ είναι κατασχέσεις μόνο της Φίλιπ Morris στο διάγραμμα αυτό. Μία λοιπόν από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ήδη είναι ότι η Φίλιπ Μόρις είναι αυτή η οποία αποφασίζει ποια ε, από τα τσιγάρα αυτά είναι αυθεντικά και ποια είναι λαθρέα και πληρώνει πρόστιμα, ή μάλλον δεν θα τα αποκαλούμε πρόστιμα, συμπληρωματικές πληρωμές εάν τα προϊόντα αυτά είναι αυθεντικά όταν κάνουμε σύγκριση των στοιχείων κατάσχεσης με τα παραποιημένα τσιγάρα, βλέπουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Για να δούμε λίγο περισσότερο τα στοιχεία της βιομηχανίας, που εδώ ε, ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο. Έχουμε στοιχεία τα οποία ε, συλλέγονται από τις άδειες συσκευασίε. Αυτά τι είναι, άδειε συσκευασίε οι οποίες έχουν πεταχθεί είτε στο δρόμο είτε σε δημόσιου. Ε, ε, καλά τους αχρήστων και ε, προσπαθούμε από εκεί και πέρα να δούμε αν είναι εγχώρια ή μη εγχώρια αυτά τα προϊόντα. Τα μη εγχώρια προϊόντα ε, θα μπορεί να είναι νόμιμα ή παράνομα. Αλλά στι άδειε συσκευασίε δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των δύο. Αν δούμε, για, βρούμε για παράδειγμα ένα πακέτο Μάλμπορο από το Λουξεμβούργο, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιο απλώ έχει κάνει αγορά στο Λουξεμβούργο νόμιμα ή αν έχει εισαχθεί παράνομα στη χώρα. Επομένως αυτά θεωρούνται ε, μη εγχώρια προϊόντα αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι νόμιμα ή παράνομα δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα παράνομα τσιγάρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ακριβή μέτρηση των ε, μη εγχώριων προϊόντων, εάν ε, γίνει κατάλληλη καταμέτρηση. Και πάλι όμω υπάρχουν αρκετέ ανησυχίε. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία μεθοδολογία. Η Japan Tobacco στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε μια μελέτη, ε, στην οποία δεν έδινε καμία μεθοδολογία. Πολλά από τα στοιχεία πλέον δημοσιεύονται απλώ μέσω δημοσιευμάτων στον τύπο και πάλι και εκεί δεν μα δίνεται καμία μεθοδολογία. Η καπνοβιομηχανία αρνείται να μα δώσει μεθοδολογία. Υπάρχει και σχετικό έγγραφο των συναδέλφων και ακόμα και στο Project Star όπου υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα αφιερωμένο στη μεθοδολογία δεν δίνονται αρκετέ λεπτομέρειε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καταλήλω τι μεθόδου. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίου ανησυχούμε και θα επανέλθω σε αυτό. Okay. Ίσως μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μας είναι ότι ε, η υπηρεσία για τις άδειες συσκευασίες τσιγάρων ε, ίσως βρίσκει απλώς αποτελέσματα τα οποία είναι ε, ε, αποτελέσματα που ευνοούν την καπνοβιομηχανία και, τις αντίστοι, και τα αντίστοιχα λόμπι. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Ε, το, στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχη υπηρεσία ε, σε αθλητικές εκδηλώσεις και σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις μαζεύει άδειες συσκευασίες. Ποιος χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευασίες συνήθως άνδρες και ποιος πηγαίνει σε αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις συνήθως άνδρες. Στην Πολωνία βρίσκουμε υψηλότερα ποσοστά ε, παρανόμων τσιγάρων από τα επίσημα στοιχεία. Ε, και μάλιστα σε μία ανεξάρτητη μελέτη που έκανε ένας συνάδελφος, ε, όταν έγινε μία έρευνα και ζητήθηκε, ε, ρωτήθηκαν οι χρήστες εάν χρησιμοποιούσαν παράνομα τσιγάρα ή αν είχαν αγοράσει τσιγάρα λαθρέα, τα ποσοστά ήταν διπλάσια από αυτά τα οποία καταγράφονται. Στη Γερμανία συστηματικά ε, δίνεται υπερβολική εκπροσώπηση κάποιων περιοχών στα σύνορα και γύρω από τις στρατιωτικές βάσεις ε, των ΗΠΑ. Και μάλιστα όταν είχαμε να έχουμε αυτές τις εκθέσεις και την αύξηση στο παράνομο εμπόριο, είχαμε ταυτόχρονα στο Ηνωμένο Βασίλειο τη συζήτηση για τις ε, απλές συσκευασίες χωρίς καμία ένδειξη. Από εκεί διαπιστώνεται ότι γίνεται αλλαγή στη μεθοδολογία ώστε να είναι παραφουσκωμένα τα στοιχεία του 2012 σε σχέση με το 2011 γιατί τότε συζητούνταν το θέμα. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα στην ε, πάνω γραμμή είναι τα στοιχεία από την ε, ε, Ένωση Καπνοβιομηχάνων του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, η έρευνα αυτή βρίσκει υψηλότερα ποσοστά από άλλες και εδώ έχουμε μια σειρά ανάμεικτες γραμμές, μία πάνω στην άλλη και εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε κυβερνητικά στοιχεία και στοιχεία της καπνοβιομηχανίας που βρίσκουν αντίστοιχα δεδομένα και πάμε και στο 2011 όπου ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή, υπάρχει μία συνεχής μείωση των ε, κρατικών στοιχείων και μειώνεται αυτό ακόμα και περισσότερο στα πιο πρόσφατα στοιχεία, αλλά η καπνοβιομηχανία έχει μία ξαφνική αύξηση. Σε μία δεν έχουμε καμία μεθοδολογία και στον άλλη έχουμε το Project Star που έχει αλλάξει τη μεθοδολογία του. Και επομένως έχουμε στοιχεία από ε, τις κυβερνήσεις που μας δείχνουν ότι έχουν πέσει τα ποσά και έχουμε και δύο ανεξάρτητες έρευνες που μας έχει δείξει ότι μειώνεται και πάλι ε, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δούμε όλα τα δημοσιεύματα στον τύπο για τη λαθρέα τσιγάρα, όλα αυτά βασίζονται σε έρευνες για άδειες συσκευασίε και διαπιστώνεται ότι έχει άρξει αύξηση μεταξύ του 2011 και του 2012 εγώ τα αναφέρω ως ε, παράνομα γιατί ε, αναφέρονται ως παράνομα στις, ε, στα δελτία τύπου αλλά είναι απλώς μία εγχώρια τσιγάρα γιατί όλα αυτά τα προσμετρούμε ως παράνομα η ε, έρευνα για τις άδειες συσκευασίες μας δείχνει ότι υπάρχει μια ξαφνική αύξηση, ενώ όλες οι επίσημες ε, έρευνες μας δείχνουν ότι υπάρχει μείωση ε, των παράνομων τσιγάρων μέχρι και το 2013 όμως, όπου φαίνεται ότι από τα κυβερνητικά στοιχεία υπάρχει μια ελαφρά αύξηση. Τώρα, δεν έχω πολλά χρόνο να επισέλθω σε λεπτομέρειες για αυτά. Εδώ έχουμε τα παράνομα μία χώρια προϊόντα, διότι προσπαθούμε με άλλους τρόπους, με άλλα δεδομένα, να προσμετρήσουμε και τη νόμιμη πτυχή όλων αυτών των ε, ε, μη εγχώριων προϊόντων. Τι κάνουμε λοιπόν, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του Project Star με τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης μελέτης η οποία δημοσιεύτηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και εκεί ζητήσαμε ε, να μας πούν εάν χρησιμοποιεί ο κόσμος λαθρέα τσιγάρα ε, και προσπαθούσαμε να έχουμε κάποια στοιχεία και βλέπουμε ότι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε ε, ε, μπορούμε να το πάρουμε και να το συγκρίνουμε με τα στοιχεία που έχουμε στο Project Star. Αν δούμε όλες τις χώρες και τις 16 χώρες που βρίσκονται σε αυτές τις δύο πηγές ε, δεδομένων, το Project Star και των εκτιμήσεων που κάναμε, κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο και από τις 16 χώρες στις 12 ε, οι εκτιμήσεις στο Project Star ήταν υψηλότερο. Τα τρία τέταρτα λοιπόν των χωρών που μπορούσαμε να συγκρίναμε είχαν υψηλότερες εκτιμήσεις του Project Star και οι χαμηλότερες εκτιμήσεις ε, ήταν σε χώρες στις οποίες υπάρχει ε, δυνατότητα αγοράς ε, στα σύνορα. Την Αυστρία, τη Γαλλία για παράδειγμα. Πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα για την έρευνα των άδειων συσκευασών, των εγχώριων και μη εγχώριων. Οι μη μπορεί να είναι νόμιμες ή παράνομες συσκευασίες. Και έχουμε αφορολόγητα τσιγάρα, τα οποία μπορεί να φέρουν τουρίστες, ε, φοιτητές, αλλοδαποί, μετανάστες ε, και φυσικά διασυνοριακές πωλήσει. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι η έρευνα για τις άδειες συσκευασίες διεξάγεται σε πόλεις, ε, όπου υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και τουριστών. Και επίσης ε, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις διασυνοριακές πωλήσει και να τις λάβουμε και αυτές υπόψη για να μπορέσουμε να έχουμε μια εκτίμηση των λαθρέων τσιγάρων. Και γίνεται μια έρευνα στα σύνορα, αλλά ε, ρωτούνται οι πολίτες μόνο για τσιγάρα τα οποία αγόρασαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους. Ε, και αυτό φυσικά δεν μας επιτρέπει να μετρήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι απλώς περνούν τα σύνορα για να αγοράσουν τσιγάρα, γιατί ζουν σε μεθοριακές περιοχές. Και τέλος ένα ακόμα πρόβλημα στο δεδομένα του Project Star είναι να καθορίσουμε κατά πόσον τα προϊόντα είναι ε, μια αυθεντική μάρκα της ε, καπνοβιομηχανίας ή κάποια απομίμηση η οποία παράγεται από την ίδια την καπνοβιομηχανία και εγώ επιμένω ότι εκεί υπάρχει διαφορά διότι καταβάλλονται πρόστιμα μόνο για τα ε, παραποιημένα προϊόντα. Τα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχουν ε, συνεχείς ενδείξεις ότι συμμετέχει η ίδια η καπνοβιομηχανία ε, στο λαθρεμπόριο τσιγάρων ε, οι συμφωνίε φαίνεται ότι δεν έχουν αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τις καπνοβιομηχανίες και συμμετέχουν ακόμα σε παράνομη διακίνηση τσιγάρων. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα στοιχεία τη καπνοβιομηχανία για τα λαθρέα τσιγάρα. Οι έρευνε ε, για τι άδειε συσκευασίε ε, υπάρχουν ενδείξει ότι χρησιμοποιούνται για να τι θέσει που υποστηρίζουν οι ομάδε πίεση. Και επίση υπάρχουν πολλά δεδομένα ναι μεν για τα παράνομα τσιγάρα από την καπνοβιομηχανία, αλλά έχουμε ελάχιστα στοιχεία από άλλες πηγές. Ενδείξεις ότι ανεβαίνουν ε, υπάρχουν μόνο από τα στοιχεία του Project Star. Αν ε, δείτε τα στοιχεία των κατασχέσεων, ε, θεωρούμε ότι υπάρχει μείωση στα λαθρέα τσιγάρα. Η απάντηση είναι γενικότερα ότι δεν ξέρουμε γιατί δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία. Και επίσης δεν μπορούμε να βασιστούμε και στα στοιχεία για τα λαθρέα τσιγάρα γιατί δεν είναι τα προσωπευτικά για αυτά που έχουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητρία Γκίλμορ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε και τα στοιχεία που παρουσιάσατε. Και είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Κυρία Γκίλμορ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς μας παρουσιάσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Έχετε και πολλά στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει, πολλές μελέτες που έχουν δημοσιεύσει οι συνάδελφοί σας σε επιστημονικά περιοδικά. Έχουν δημοσιευτεί λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω στις ε, έρευνές σας και δεδομένου του γεγονότος ότι έχετε βαθιά γνώση του αντικειμένου σας έχουν Σας έχουν προσεγγίσει, λοιπόν, ποτέ ε, αρχές κρατών μελών και αν ποιες δεδομένων όσων μας είπατε ότι εμπλέκεται η καπνοβιομηχανία στα, στο διακίνηση παράνομων τσιγάρων. Έχετε συζητήσει ποτέ με την Γενική Διεύθυνση Τάξουτ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον ε, Επίτροπο για θέματα απάτηση το επιτελείο του. Είχατε επαφές με τον Όλαφ και εάν ναι, τι έγινε και ποιε αντιδράσεις ε, υπήρξαν από τις ε, πληροφορίες που τους δώσατε και έπειτα έχετε κάποιες πληροφορίες να μας πείτε σχετικά με το τι κάνει ο Επίτροπος ΕΣΕΜΕΤΑ για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Υπήρξε μία ανακοίνωση τον Αύγουστο του 2013 και μία μελέτη που δημοσιεύθηκε. Ε, εσείς συμμετείχατε στην ε, σύνταξη αυτής της ανακοίνωσης. Αυτά που μας είπατε είναι πραγματικά σοκαριστικά. Και σίγουρα αυτά που λέτε δεν τα ακούει κανείς ευχάριστα. Και ιδιαίτερα η καπνοβιομηχανία, η οποία δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνεί και 100% με όσα είπατε. Λοιπόν, σας έχουν προσεγγίσει ποτέ από την καπνοβιομηχανία. Έχει υπάρξει διάλογος ή κάποια διαφωνία. Και τι διδάγματα έχετε αντλήσει από αυτό. Πώς μπορούμε δηλαδή να χειριστούμε αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκρέσλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Δεν μπορούσα να βρω την παρουσίαση στο ενημερωτικό αυτό φυλάδιο, αλλά θα την ψάξω. Νομίζω πως έχει διανεμηθεί κιόλα. Εδώ είναι. Δεν την είδα. Όλο αυτό το θέμα με την έκθεση για το project STAR και για την αξιοπιστία των δεδομένων είναι κάτι ανησυχητικό. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μας συμβουλεύετε και μετά από όλα όσα είδαμε και μετά από τις έρευνες των άδειων πακέτων υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα και στο σύστημα επισήμανσης. Γι' αυτό λοιπόν τι συμβουλές θα έχετε εσείς να δώσετε στους συναδέλφους και σχετικά με τις ενέργειες του Όλαφ επίσης. Ευχαριστώ. Προτείνω να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερες ερωτήσεις. Ο κύριος Σόραν Χίτεγκάρτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Μία ερώτηση έχω. Δεν ξέρω αν ταιριάζει ε, με αυτά που μας είπατε, με τις αρμοδιότητές σας. Όμως, θα ήθελα να μάθω τα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν από την καπνοβιομηχανία. Πόσο διαφέρουν από τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου που έχετε εσείς, τι γίνεται με την καπνοβιομηχανία Και ποιους λόγους έχει για να κάνει όλα αυτά, μας είπατε. Ένας ε, από τους λόγους που αναφέρεται ήταν η μεγιστοποίηση των κερδών τους σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η μισθή είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Όμως, έχετε την εντύπωση ότι η καπνοβιομηχανία έχει μεταφέρει τις μονάδες παραγωγής σε χώρες με λιγότερους ελέγχους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκίλμορ, μπορείτε να Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν ότι για την πρώτη ερώτηση έχω εργαστεί με τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες. Δεν συνεργάστηκα όμως με τον Όλαφ, δεν με πλησίασε ο Όλαφ. Αντίθετα, η αρμόδια υπηρεσία για τα έσοδα του κράτους του, της Μεγάλης Βρετανίας με την οποία συνεργάστηκα, με την DG7, για το πρόγραμμα το οποίο αναφέρθηκε. Επίσης, όσον αφορά την έρευνα, βεβαίως ε, εμείς ε, δώσαμε στη διάθεση του Όλαφ κάποια από τα στοιχεία. Είχαμε πολλές ε, συναντήσεις και αλληλογραφία με την καπνοβιομηχανία. Τα κύρια στοιχεία που πήρα ήταν όσον αφορά τις κατασχέσεις και τα ποσά των κατασχέσεων. Προσπάθησα λοιπόν εγώ να βγάλω άκρη παίρνοντας τα στοιχεία του προγράμματος STAR, κάνοντας μία διαίρεση με το ποσό των κατασχέσεων, τα στοιχεία από το STAR, αλλά και όλα αυτά που είχα από τη Philip Morris και έφτασα σε ένα τελικό ποσοστό 9 cents του ευρώ για περίπου 100 τεμάχια τσιγάρων. Αυτό ήταν το τελικό ποσό που είδα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τα στοιχεία που έχω για τις κατασχέσεις, σε αυτό το αποτέλεσμα έφτασα. Άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ΣΤΑΡ. Κοιτάξτε, το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το πρόγραμμα είναι καλό. Ουσιαστικά είναι στοιχεία των 27 κρατών μελών με διαφορετικές πηγές βεβαίω στοιχείων. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της παράνομης διακίνησης τσιγάρων στηριχτήκαμε σε αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Κάποια από αυτά βεβαίως ε, εδώ, κάποιες πηγές ε, μπορεί να έχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα STAR, σαφώς και δεν θα πρέπει να καθοδηγείται από την καπνοβιομηχανία, από μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία και να υπάρχει και περισσότερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα. Άλλη ερώτηση έλεγχος των καπνοβιομηχανιών και ο έλεγχος ε, πόσο διαφέρει στα διάφορα κράτη-μέλη, αν υπάρχει πιο χαλαρός έλεγχος σε κάποια κράτη-μέλη. Ναι, σίγουρα είναι πιο φτηνή η παραγωγή τσιγάρων στην Λευκορωσία, στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Η έλεγχη είναι πιο χαλαρή και δυστυχώς η διαφθορά είναι πιο σημαντική. Αυτό διευκολύνει την δραστηριότητα την παράνομη. Αυτό νομίζω ότι ολοκληρώνει και τις απαντήσεις μου. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μία ερώτηση για σας. Ίσως δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Αλλά στις ε, έρευνές σας στην επιστημονική σας έρευνα διαπιστώσατε λόγους για τους οποίους η καπνοβιομηχανία στοχεύει τόσο πολύ στο παραεμπόριο τσιγάρων. Κάποιος άλλος νομίζω όμως θέλει να πάρει το λόγο. Ναι. Μπορείτε να πείτε και ποιος είστε αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Adrian Welsh και είμαι επικεφαλής ε, των διοικητικών ε, αρχών για τα προϊόντα καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να σας πω ότι το Σεπτέμβριο του 2010 υπογράψαμε μια συμφωνία με την καπνοβιομηχανία. Προαιρετική ήταν αυτή η συμφωνία και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Γκίλμορ όσον αφορά την αξία αυτών των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και είμαστε δεσμευμένοι και όπως είπε και η κυρία Γκίλμορ δίνοντας ε, την, ε, σαν παράδειγμα τη μάρκα Classic που παρασκευάζονται στην Ουκρανία. Η μάρκα αυτή είναι πολύ σημαντική για μας και την παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, διότι παρακολουθούμε βάσει της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντοπίσαμε και αν κοιτάξει κανείς ε, αυτά που αναφέρει το σχέδιο STAR όταν αναφέρεται για αυτά τα παράνομα άσπρα τσιγάρα, δηλαδή τσιγάρα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι παραποιημένα αλλά εν πάση περιπτώσει διακινούνται μέσω του λαθρέου δικτύου. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι κατασχέσεις τέτοιων τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσό τέτοιων τσιγάρων το οποίο όμως σε σχέση με τα παραποιημένα τσιγάρα είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι περίπου 21 εκατομμύρια τσιγάρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και παρακαλώ πολύ σημειώστε το. Εμείς πραγματικά θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο και θεωρούμε ότι αυτές οι παράνομες δραστηριότητες οι οποίες αποδυναμώνουν την, ε, ε, τον τομέα των γνήσιων τσιγάρων και ιδιαίτερα όσον αφορά τη μάρκα Classics και την ε, παρασκευή από την Ουκρανία τα στοιχεία που διαθέτουμε που είναι του Οκτωβρίου 2012 δείχνουν ότι έχει σταματήσει τελείως η παραγωγή αυτών των τσιγάρων Classics και τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ότι σταμάτησε τελείως η παραγωγή τους ήδη από τον Ιούνιο του 2013. Αυτά τα τσιγάρα που βλέπουμε να εισάγονται είναι παραποιημένα τσιγάρα. Πρόεδρος. Η Ίνκε Γκρέσλα έχει ακόμα μια ερώτηση. Σας ζήτησα να πάρετε θέση και να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο για το σύστημα track and trace, ανείχνευσης παρακολούθησης και αν έχετε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα λαθρέα τσιγάρα, τα παραποιημένα τσιγάρα. Και μια άλλη ερώτηση που ήθελα να μου απαντήσετε. Ποια είναι η άποψή σας, πώς βλέπετε εσείς αυτήν την συμφωνία Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά επιτρέπει κάποια πράγματα υπό κάποιες ε, βεβαίως νομικές ε, διατάξεις και προϋποθέσεις, όπως παραδείγματο χάρη την επιβολή προστήμων. Εσείς ε, πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τη στάση της καπνοβιομηχανίας. Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολλές ε, συνεδριάσεις και συναντήσεις που είχατε με τους εκπροσώπους της καπνοβιομηχανίας, σε τι συνολικό αποτέλεσμα σας οδήγησαν όσον αφορά τη στάση της καπνοβιομηχανίας. Πρώτη ερώτηση. Γιατί υπάρχει λαθρέα διάθεση τσιγάρων. Καταρχήν, φυσικά και η καταπολέμηση και η δίωξη είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς και η διάθεση παράνομων τσιγάρων βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή. Γι' αυτό και αγοράζονται, γι' αυτό και διατίθενται. Και έτσι κι αλλιώ, από τη στιγμή που είναι παραποιημένα και λαθρέα τα τσιγάρα, προσπαθούν να τα διοχετεύουν σε μεγάλε ποσότητε μέσω αυτών των δικτύων. Οπωσδήποτε όμως, οι καταναλωτές εδώ και εδώ απαντώ στη δεύτερη ερώτηση είναι οι νέοι καταναλωτές, οι οποίοι σαφώς και προσπαθούν να αγοράσουν τσιγάρα σε χαμηλότερες τιμές. Τώρα, όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, είσοδος της αγοράς και οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάποια στιγμή στην αρχή της δεκαετίας του 90 οι αγορές ήταν κλειστές για κάποια προϊόντα, για κάποιες αγορές, για κάποιες χώρες, οι καπνοβιομηχανίες ξεκίνησαν με λαθρέο τρόπο τη διάθεση γνήσιων τσιγάρων, γνήσιων προϊόντων. Αυτές οι χώρες ουσιαστικά παραμένουν και σήμερα οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό λαθρεμπορίου τσιγάρων. Οι καπνοβιομηχανίες χρησιμοποιούν αυτό το λαθρεμπόριο τσιγάρων σαν ένα επιχείρημα για την στρατηγική τους. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, σαν αποτέλεσμα των ερευνών στη Μεγάλη Βρετανία που βασίζεται στα άδεια πακέτα που μαζεύουμε, δείχνουν ακριβώς αυτό ότι ουσιαστικά εδώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το λαθρέο εμπόριο μπορούμε να πούμε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας. Τώρα, στο ερώτημα για την μάρκα Classics από την Ουκρανία και γιατί έφτανε και πουλιόταν μέχρι και στην Ευρώπη. Μου λέτε ότι δεν ήταν παραποιημένο και η απάντησή μου είναι ναι, αλλά έτσι όπως είναι αυτό το προϊόν γιατί κάποιος να το παραποιήσει. Το θέμα των illicit white, των ε, παράνομων λευκών τσιγάρων. Εδώ και χρόνια πολλούνται αυτά τα τσιγάρα και το ποσοστό τους φτάνει το 7% των πολλούμενων τσιγάρων στην αγορά. Το τελευταίο σημείο, κοιτάξτε δεν είμαι εμπειρογνώμονας για το σύστημα track and trace, θα απαντήσουν οι ειδικοί σε αυτή την ερώτηση που είναι εδώ μαζί μου. Αλλά στην άλλη σας ερώτηση που αφορά την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Τα καλά αυτής της συμφωνίας είναι πρώτον ότι η καμπρομιομηχανία είχε πολύ καλύτερη γνώση των δεδομένων της ε, ρυθμιστικής ε, δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για τον τομέα της καπνοβιομηχανίας. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι η συμμετοχή της καπνοβιομηχανίας σε όλες αυτές τις ρυθμιστικές δραστηριότητες ήταν σημαντική. Υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με την Όλαφ, ανεπαρκής κατά την άποψή μου. Η συμμετοχή δηλαδή της καπνοβιομηχανίας δεν είναι επαρκής σε όλη αυτή τη στρατηγική. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ίσως προβληματικό να συνεργαζόμαστε τόσο πολύ με την καπνοβιομηχανία η οποία ουσιαστικά είναι ε, τμήμα του προβλήματος που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική που βασίζεται στην αποτροπή δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Πρόεδρος. Μία ερώτηση μόνο ακόμα για την κυρία Γκίλμορ. Δεν ξέρω αν αυτή η ερώτηση ουσιαστικά πρέπει να απευθυνθεί σε εσά ή σε κάποιον άλλον αργότερα. Μιλήσατε για το θέμα του λαθρεμπορίου τσουγάρων. Εγώ δεν καπνίζω, δεν είμαι καπνίστρια. Αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η διερεύνηση που έχει γίνει για τις άλλες οδούς ε, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Γιατί παραδείγματο χάρη υπάρχουν ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Υπάρχουν φυσικά και χώρες στις οποίες ξέρουμε ότι εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη στη χώρα μου την Αυστρία, με παράνομο τρόπο από πολλά διαφορετικά δίκτυα και ότι κάποια τσιγάρα περνάνε από το λαθρεμπόριο στο επίσημο εμπόριο, παράνομα τσιγάρα αγοράζονται και καπνίζονται από τον Ευρωπαίο καταναλωτή χωρίς να το γνωρίζει. Γιατί διακινούνται από το επίσημο δίκτυο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Κυρία Γκίλμορ, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή και βεβαίως ενδεχομένως και άλλοι εμπειρογνώμονες αργότερα μπορούν να επανέλθουν σε αυτές τις ερωτήσεις και να απαντήσουν. Κυρία Γκίλμορ, θέλετε να απαντήσετε, αν, εάν θέλετε. Πολύ Θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι πολύ περίπλοκο. Έχουμε διάφορα και προσπαθούσα να τα αντιμετωπίσω. Έχουμε τα παράνομα λευκά, τα οποία παράγονται νομίμως αλλά διοχετεύονται στην παράνομη αγορά. Υπάρχουν τα παραποιημένα, απομιμήσεις δηλαδή και μετά υπάρχουν οι αυθεντικές μάρκες στις καπνοβιομηχανίες που ε, παράγονται ε, σε πολύ μεγαλύτερο ε, όγκο στην αγορά γνωρίζοντας ότι θα διακινηθούν στη συνέχεια παρανόμως κάποια από αυτά στα σύνορα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αν καπνίζουν παράνομα ή νόμιμα τσιγάρα. Αυτό νομίζω απαντά στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκίλμορ για την συνεισφορά σας. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον Χάουαρτ Πιού, από την Ευρωπόλ. Um, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για την πρόσκληση για να έρθω εδώ να σας μιλήσω λίγο για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. Ε, ήμουνα σε θέματα ποινική δίωξης ε, στο Τελωνείο. Ε, ήμουνα και σύνδεσμος ε, στη χώρα μου και τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζομαι για την Ευρωπόλ ως... Ε, ε, επικεφαλής αναλυτής. Ε, Κεντρώνομαι ε, στα, στις αιστείες τσιγάρων. Έχω μια ομάδα αναλυτών που προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση του οργανωμένου εγκλήματος με τη λαθρέα διακίνηση τσιγάρων. Τι κάνει η Europol λοιπόν. Η Europol είναι οργανισμός εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επικεντρωνόμαστε σε θέματα ποινική ε, δίωξης, ε, συλλέγουμε, αναλύουμε και διαδίδουμε πληροφορίες στις υπόλοιπες μονάδες επιβολής του νόμου. Και ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουμε είναι η διευκόλυνση ανταλλαγή πληροφοριών με δύο τρόπου. Ε, πρώτον, μέσω ενό ασφαλού συστήματο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ΣΥΕΝ, που έχει πρόσβαση όχι μόνο σε ανθρώπου στο ίδιο κτίριο, αλλά και σε άλλου οργανισμού ε, στα κράτη-μέλη και στι αρμόδιε αρχέ με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Και υπάρχει και ένας αριθμός ε, συνδέσμων που εδρεύουν στην Ευρωπόλ και ε, δρούν ο σύνδεσμος και δίωδος ε, στις εθνικές υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Καθημερινά υποστηρίζουμε επιχειρησιακά και στρατηγικά μέσω ανάλυσης τις έρευνες των οργανισμών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών και θέλουμε να καλύψουμε σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα και τρομοκρατία. Αυτή είναι η εντολή μας και χρειαζόμαστε πάντα δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη ε, για να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Η έδρα μας είναι στη Χάγη, εδώ βλέπετε το κτίριό μας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα αμάλγαμα αναλυτών, ειδικών και αξιωματικών συνδέσμων και όλα αυτά ε, σε στενή επαφή με τις ε, ε, ε, υπηρεσίε τη αρμόδια των κρατών μελών, αλλά και με χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από του βασικού αριθμού που έχουμε είναι το 71. Έχουμε 71 οργανισμού ε, που συνεργάζονται με την Ευρωπόλ και στο παρελθόν θεωρούσαν ότι ήμασταν απλώ αστυνομική υπηρεσία, αλλά δεν ισχύει αυτό. Έχουμε 145 αξιωματικού συνδέσμου που εδρεύουν στην Ευρωπόλ και αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμό στου 180 περίπου. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στον κόσμο που ε, να στεγάζουν τόσους πολλούς ε, αξιωματικούς ε, που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου. Ε, η ομάδα εργασίας είναι η αγγλική και εγώ πολύ σύντομα μπορώ να έρθω σε επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες για να δούμε ποιος χρειάζεται τι για να συνεχίσει η επιτήρηση και ποιος έχει πόρους για να συνεχίσει αυτή την έρευνα αν απαιτείται. Europol η Europol έχει μία προσέγγιση πολλαπλών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Στο κτίριο αυτό έχουμε ε, αστυνομία, τελωνία, χωροφυλακή, ε, ε, τελωνιακούς υπαλλήλους, υπηρεσία μετανάστευσης και πολλούς άλλους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τη μορφή των εγκλημάτων που ερευνούμε. Στην Europol έχουμε τα 28 κράτη-μέλη Έχουμε και 13 τρίτα μέρη ε, που συμμετέχουν αξιωματικού συνδέσμους και μπορούμε να έχουμε μόνο 12, ε, μάλλον συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχουμε 12 επιχειρησιακές συμφωνίες με άλλες χώρες και έχουμε ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές και τους αρμόδιους οργανισμούς και έχουμε και 20 στρατηγικές συμφωνίες με χώρες και οργανώσεις που μας επιτρέπουν να ανταλλάσσουμε τάσεις, τάσεις, operandi και τέτοιες λεπτομέρειες, χωρίς βέβαια να γίνεται ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Η ομάδα μου ε, συνεργάζεται με τρεις άλλες ομάδες. Εμείς είμαστε ε, το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ε, ε, υπάρχει επίσης ε, μία ομάδα που ασχολείται με την απάτη ΦΠΑ μία άλλη η οποία ασχολείται με τις ομάδες ε, οι οποίες ε, αποτελούν εστίες ε, και έχουμε και μία τέταρτη ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε και όλοι αυτοί προσπαθούμε να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση του εγκλήματος, διασταυρώνουμε στοιχεία με τα διάφορα αρμόδια τμήματα, εμείς επικεντρωνόμαστε στον καπνό και υπάρχουν και 23 άλλες ομάδες. Όλα τα στοιχεία τα οποία εξεργάζεται η Europol σήμερα τα διασταυρώνουμε με άλλα στοιχεία και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλυση. Και προσπαθούμε να βρούμε σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, αριθμητικών στοιχείων, επιχειρήσεων, πινακίδων αυτοκινήτων, μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, διαφορετικών υπηρεσιών και διαφορετικών περιοχών. Το λαθρεμπόριο καπνού ε, έχω πάρει από την έκθεση Project Star ε, και ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντική η συμμετοχή της Ευρωπόλη είναι γιατί η απώλεια εσόδων για τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εκτιμάται το 2012 στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για ανθρώπους οι οποίοι ε, διακινούν λαθρέα ε, προϊόντα καπνού ή παράγουν ε, λαθρέα τσιγάρα. Αυτό επιτρέπει σε εγκληματίες ε, να έχουν έσοδα για να ασχολούνται και με άλλους τομείς του οργανωμένου εγκλήματος και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση με ναρκωτικά, όπλα, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και αντίστοιχες μορφές αδικημάτων. Ε, ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάλυση είναι ε, διότι ε, μόνο 2% από τα 500 εκατομμύρια εμπεριβηματοκιβώτια τα οποία διακινούνται ετησίως επιθεωρούνται. Αυτά είναι στοιχεία από το UN ODC. Και προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τους κακούς, όχι μόνο να στοχεύσουμε στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. So my team itself, what we aim to do το τμήμα μου προσπαθεί να στοχεύσει στις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που συμμετέχουν στην παράνομη ε, ε, παρασκευή και διακίνηση προϊόντων καπνού. Ε, προσπαθούμε να περάσουμε απευθείας από τους οδηγούς και αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν τσιγάρα στα ανώτερα στελέχη για να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης ε, έχουμε τη λεγόμενη ε, πολιτική επιβολή του νόμου, έχουμε πολύ ε, τομιακές πλατφόρμες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι επικεφαλής για τα εμπορευματοκιβώτια που είναι ο τελευταίος κύκλος πολιτικής και θα είμαι και επικεφαλής ε, για τα θέματα των φόρων ειδικής κατανάλωσης τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να δούμε ε, όχι μόνο τον καπνό, αλλά όλα τα ε, θέματα απάτης φόρων ειδική κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα τα ενοπνευματόδη και οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα κατά την άποψή μας που βοηθά στην επιβολή του νόμου είναι οι πληροφορίες ε, και η αστυνόμευση μέσω των πληροφοριών που συλλέγονται. Προσπαθούμε να έχουμε πληροφορίες για το εμπόριο, για την ιδιωτική βιομηχανία και τις ανοιχτέ πηγές και προσπαθούμε να δώσουμε μια ε, καλύτερη εικόνα του προβλήματος. Και έτσι μπορούν οι ομάδες επιβολής του νόμου να χρησιμοποιήσουν τους περιορισμένου πόρου που έχουν για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πλήττει την κοινωνία μα. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το πρόβλημα ε, και μπορούμε ε, να χρηματοδοτήσουμε επιχειρησιακές συσκέψεις, ε, να τις υποστηρίξουμε και από εκεί και πέρα να υπάρξει και κάποια συνεχής αναλυτική υποστήριξη. Για τον ε, καπνό έχουμε 26 εστίες ε, στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Ε, προσφάτως εντάχθηκε και το Βέλγιο, μόλις πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 6 εταίρους από περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμαστε και με τη Eurojust για παράδειγμα στενά που μας δίνουν Είναι σε θέματα δικαιοδοσίας σε διασυνοριακά προβλήματα. Επίσης, προσφάτως ε, ξεκίνησε και μία συνεργασία με την FDA των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Food and Drug Administration και υπάρχει συνεργασία με την Olaf. θα ήθελα να σας επισημαίνω τέσσερις τομείς ε, του παράνομης διακίνησης καπνού οι οποίοι μας απασχολούν. Παραδοσιακά εξετάζουμε τις απομιμήσεις τσιγάρων, ε, ε, τσιγάρα τα οποία μοιάζουν με αυθεντικά προϊόντα, συνήθως προέρχονται από την Κίνα, προσφάτως όμως ε, ε, και πιο κοντά. Φαίνεται ότι έχει ε, γίνει πιο σύντομη η αλυσίδα εφοδιασμού και αυτό δίνει τη δυνατότητα ίσως παρέμβασης. Αν έχουμε ένα εμπορευματοκιβώτιο που έρχεται από την Κίνα, έχεις δύο με τρεις εβδομάδες να το εξετάσεις. Αλλά είναι ένα φορτηγό το οποίο έρχεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Φθηνά λευκά τσιγάρα κυρίως παράγονται σε χώρες όπως η Μέση Ανατολή ε, και αποτελούν πλέον ουσιαστικό πρόβλημα. Μοιάζουν με γνωστές μάρκες, αλλά είναι σχεδιασμένα απλώς να μοιάζουν και ε, ίσως έτσι μπορούν να ξεφύγουν και από κάποιες πλευρές ε, παραβίασης αγοράς και παρανομίας. Παράνομα εργοστάσια παραγωγής καπνού. Εδώ έχουμε τεράστια ζημία Έχουμε 600-700 χιλιάδες ευρώ αξία, πολλές φορές η παραγωγή είναι μυστική και παράγονται ε, εμπορευματοκιβώτια και αποστολές κατά παραγγελία. Απλώς ε, γίνεται ε, εισαγωγή και χρησιμοποιούν όμως ε, ε, και διάφορα συστατικά τα οποία είναι παγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρασκευάσουν τα τσιγάρα τους. Και Πρόσφατα ε, μας επέστησαν την προσοχή αρκετά κράτη-μέλη το ε, ότι μπορεί να γίνεται και παράνομη χρήση του συστήματος ελέγχου ε, και διακίνησης σε προϊόντα ε, που υπόκειται σε φοροειδικής κατανάλωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα καθεστώτα. αν όμως στη συνέχεια δίνει κάποιος, κάνει κάποιος μία μεταφορά σε κάποια περιοχή στην οποία δεν είναι συνήθις περιοχή ελέγχου, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να διαφύγει τον έλεγχο και να μην καταβληθεί φόρος. Έτσι έχουμε παράνομη διακίνηση. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να σας εξηγήσουμε λίγο πιο απτά τα πράγματα Υπήρχε μία υπόθεση η οποία προσήχθη στο δικαστήριο ε, για τελωνία. Η Europol δεν είχε εκτελεστική εξουσία. Εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε, αλλά αν μας ζητηθεί να ε, συνδράμουμε ένα κράτος μέλος, μπορούμε να μεταβούμε στο κράτος μέλος και υπήρχε και ε, στενή συνεργασία με τη Eurojust. Υπήρχε μια ομάδα η οποία διακινούσε τσιγάρα από την Ουκρανία στη Γαλλία. Οι Γάλλοι έκαναν μια κατάσχεση της τάξης των 7 εκατομμυρίων, μεγάλο ποσό για μια κατάσχεση, αλλά δεν ήταν τόσο ουσιαστικά. Κατάφεραν όμως να το συνθέσουν με άλλες δύο μεταφορές και εδώ συμμετέχουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να συγκεντρωθούν πληροφορίες, να δούμε ποιες ε, ε, ε, επιχειρήσεις εμπλέκονται και να δούμε και τι μπορούμε να συνδυάσουμε με τα νέα στοιχεία που συλλέγουν οι Γάλλοι. Το 2011 με δύο ε, ημέρες δράσης και κάποια κράτη-μέλη προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε μια δράση και είχαμε και ένα κινητό γραφείο. Ουσιαστικά είναι ένας ε, φορητός υπολογιστής ο οποίος μπορεί να συνδεθεί ε, απομακρυσμένα με τη βάση δεδομένων της Europol. Μέσω αυτού λοιπόν του τμήματος εργαστήκαμε με 150 ε, αξιωματικούς, ε, αστυνομία, τελωνία και δικαστικούς, οι οποίοι έδρασαν επιτόπου, έκαναν συλλήψεις, ε, έρευνες κατοίκων και έγιναν και δύο εκδόσεις. Ε, υπήρχαν αρκετές ε, συσκευές οι οποίες κατασχέθηκαν και μπορέσαμε να δώσουμε και στοιχεία για, την, για τις συσκευές αυτές μέσω της σήμανσης και επίσης μπορέσαμε να παρέχουμε και αναλυτική υποστήριξη ευθύ εξ αρχή, κάτι το οποίο μα βοήθησε και η Eurojust να κάνουμε. Ο λόγος για τον οποίο σας τα λέω αυτά είναι γιατί τον Αύγουστο οι Γάλλοι καταδίκασαν ε, ε, σε 10 χρόνια τον επικεφαλής ε, και τον δεύτερο τη τάξη σε 7 χρόνια για λαθρεμπόριο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα για τους Γάλλους και είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε να βοηθήσουμε. Και είναι ένα από τα καλύτερα ρεκόρ τα οποία έχουμε θέσει για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή υπόθεση την οποία ε, διεξήγαγαν πάρα πολύ καλά οι Γάλλοι σε συνεργασία με όλους εμάς. Αυτή τη βοήθεια μπορεί να παράσχει η Europol, ε, μπορούμε να έχουμε βοήθεια μέσω πληροφοριών, παρέμβαση, συντονισμό, αλλά όταν οι ύποπτοι ε, προσήχθησαν στο δικαστήριο, ο ένας εξ αυτών είπε ότι επισκέφθηκε το Ντουμπάι με την οικογένειά του και ήταν εκεί σε διακοπές, αλλά όταν δώσαμε εμείς τα στοιχεία από τη σήμανση που είχαμε, φωτογραφίες ε, και πού είχε βρεθεί και πού τον είχαμε εντοπίσει, μπορέσαμε να διαψεύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία διότι τον είχαμε ε, φωτογραφία σε εργοστάσια όπου έκανε έλεγχο των προϊόντων τα οποία θα διακινούσε ελαθρέα και φυσικά έτσι ε, ε, Διαψεύθηκε και όλη η υπεράσπιση του στο δικαστήριο και μπόρεσε να καταδικαστεί. Μια τελευταία διαφάνεια λοιπόν για το τι άλλο κάνουμε. Εδώ έχουμε ένα κινητό γραφείο, όπως σας είπα είναι απλώς ένας φορητός υπολογιστές ε, και χρησιμοποιούμε ε, και το UFED που είναι τα αρχικά για το Universal Forensic Extraction Device μοιάζει με κινητό τηλέφωνο και είναι μια συσκευή η οποία συλλέγει πληροφορίες από τα κινητά τηλέφωνα. Για παράδειγμα, αν κάποιος ε, σταματήσει στα σύνορα έναν οδηγό ο οποίος ε, έχει ένα φορτηγό γεμάτο παράνομα λαθρέα τσιγάρα μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες από το κινητό του τηλέφωνο και να μιλήσουμε με τους ερευνητές και να τους επισημάνουμε κάποιους τομείς τους οποίους δεν έχουν ψάξει ακόμα. Όπως σας είπα, προσπαθούμε να λάβουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ε, έχουμε ένα πρόγραμμα ε, ανοιχτής ε, πηγής πληροφοριών που προσπαθεί να αναλύσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν μας έχουν ε, ε, δοθεί εμάς μέσω καταγγελίας αλλά έχουν δοθεί σε κάποιες άλλες ανοιχτές πηγές και προσπαθούμε να συλλέξουμε πληροφορίες μέσω του ιδιωτικού κλάδου που μας βοηθά επίσης εμπορικά στοιχεία και φυσικά ομάδες επιβολής του νόμου και προσπαθούμε από εκεί και πέρα να δώσουμε την καλύτερη εικόνα σε όλους τους συνεργάτες μας επιτόπου. Όπως σας διευκρίνησα, προσπαθούμε να ε, έχουμε ως στόχο το οργανωμένο έγκλημα. Αν μπορούμε όμως να ευθαρρύνουμε να γίνεται και οικονομική έρευνα παραλλήλου, τότε ε, θεωρούμε ότι μόνο ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε, γιατί ο μόνος λόγος για τον οποίο δραστηριοποιούνται αυτές οι ομάδες είναι για κέρδος. Και ε, συνεργαζόμαστε με τους ερευνητές και ανακριτές ε, και ε, υπάρχει ε, μια γραμματεία την οποία στεγάζουμε εμείς για τη συνεργασία αυτή. Ολοκληρώνοντας, ελπίζω αυτά να σας διευκρινίζει λίγο το ρόλο της Europol και πόσο σημαντικό ρόλο έχει η ανάλυση και η πληροφορία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μίλησα για 15 λεπτά, αλλά είναι ευπρόσδεκτοι όλοι ε, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού να έρθουν στη Europol, να δείτε λίγο καλύτερα πώς κάνουμε τα πράγματα, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη εικόνα και υπάρχουν και κάποιες ε, πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη που είναι ευπρόσδεκτες διότι ε, προσπαθούμε να ε, στοχεύσουμε σε οικονομικά εγκλήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπάρχει στενή συνεργασία σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η συνεργασία είναι ζωτικό τμήμα τόσο κάνουμε και θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία είναι θετική. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου θέσετε. Thank you Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πιού για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Τώρα, ανοίγω τη συζήτηση. Μπάρτ, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ήταν πραγματικά τα κάρτες ενή παράθεση των γεγονότων. Τώρα μας μιλάτε για το παράνομο εμπόριο καπνού και μας αναφέρατε τέσσερα διαφορετικά είδη, τα ε, παραποιημένα τσιγάρα, τα ε, λευκά τσιγάρα, τα παράνομα εργοστάσια παραγωγής ε, καπνού σε ευρωπαϊκή επικράτεια και το σύστημα διακίνησης και ελέγχου προϊόντων που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και αναφέρατε επίσης ότι αυτοί είναι οι λόγοι για την μείωση των κατασχέσεων. Θα μπορούσατε να μας αναπτύξετε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο, διότι φυσικά αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με την νομοθεσία και μια και εμείς ασχολούμαστε με αυτό, θα ήταν πολύ χρήσιμο και για την επόμενη ε, θητεία να προσελκύσουμε τον ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτών. Σας ευχαριστώ. Κρέσλε. Μάλιστα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι η συνεργασία με τον Όλαφ. Μας είπατε ότι όντω υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες, κάποιες συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό και έπειτα πώς ε, εκτιμάτε εσείς τις αρμοδιότητες ε, του Όλαφ. Θεωρείτε πως ε, χρειάζεται κάποια αναδιάρθρωση ή θεωρείτε πως υπάρχουν αδυναμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα που ασχολείται με τα τσιγάρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σεντερκάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό με την προηγούμενη ερώτησή μου. Έχετε υπόψη τους ε, ελέγχους στα διάφορα Υπάρχουν διαφορές και αυτές οι διαφορές έχουν κάποια επιρροή στους ε, νόμιμους παραγωγούς καπνού, προϊόντων καπνού. Έχει κάποιες επιπτώσεις, ο έλεγχος επιτρέπει να διαφύγουν προς τις ε, μη νόμιμες οδούς οι παραγωγές. Έχει κάποια σχέση αυτό με τη μεταφορά των ε, μονάδων παραγωγής σε χώρες με λιγότερους ελέγχους. Έχετε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες ή είναι κασίες αυτά που μας λέτε βασμένες σε στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις από συναδέλφους, πολύ ενδιαφέρουσες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Μάλιστα. Πρώτη ερώτηση σχετικά με το σύστημα διακίνησης και ελέγχου προϊόντων που υπάρχουν σε φορούς κατανάλωσης. Υπάρχει ένα περιθώριο λοιπόν για αυτό. Υπάρχει ένα σύστημα, δεν είναι ακριβώς track and trace, αλλά μπορούμε να δούμε πότε εισάγεται κάτι. Όταν έχω κάνω μια εισαγωγή, καταχωρώ τι ακριβώς έχει φτάσει στην αποθήκη μου και πού πηγαίνει. Και Μπορούμε λοιπόν εμείς να μπούμε σε αυτό το σύστημα και να δούμε εάν δεν έχουν καταβληθεί αυτοί οι φόροι κατανάλωσης. Έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις ε, οργανωμένου εγκλήματος όπου έχουμε παρισφρήσει στα δίκτυα αυτά και έχουμε παρατηρήσει αυτές ε, τις ε, ενέργειες. Επίσης, Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται διαφορετικά από το κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις και υπάρχουν και διαφορές στην συλλογή δεδομένων και στον αριθμό των δεδομένων που συλλέγονται, κάτι που δυσχεραίνει όντω το έργο των αρχών επιβολής του νόμου. Τώρα, όσον αφορά τον Όλαφ, ε, δεν υπάρχει ανάγκη για ε, υπογραφή επιχειρησιακή ε, συμφωνία για να συνεργαστούμε. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου, υπάρχει νομική οδό στην οποία ακολουθούμε. Αυτό που έγινε ήταν στα πλαίσια του Project Impact της πειθαρχικής πλατφόρμας καταπολέμησης του εγκλήματος. Η Όλαφ λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος στο σύστημα διακίνησης και ελέγχου αυτό και συμφώνησε να συνεργαστεί με αυτά τα σημεία εστίασης. Έγινε μία πρώτη προσέγγιση τον Δεκέμβριο, έγινε μία μελέτη η οποία εστάλει τον Δεκέμβρη Ε, ζητήθηκε από τον Όλεφ να απαντήσει για το αν θα ήθελε να συνεισφέρει σε αυτήν την στρατηγική και τι πόρους μπορεί να διαθέσει. Αυτή λοιπόν η μελέτη διανεμήθηκε στα μέλη της ομάδας και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα υπάρξει και αυτή η επίσημη συνεργασία θα επιτρέψει την επίσημη ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων και θα μπορέσουμε ως εκ τούτου να συνεργαστούμε πολύ στενότερα. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες αμοιβαίας συνεργασίας, είχαν πολλές επιχειρήσεις τις οποίες συνεργάστηκαν. Εμείς συνεργαστήκαμε στενά, ήταν καλή η συνεργασία μας. Πολλές φορές ε, χρησιμοποίησαμε αυτό το κινητό γραφείο σε επιτόπιες επιχειρήσεις, σε μονάδες ελέγχου, οι οποίες είχαν οργανωθεί από τον Όλαφ. Αφορούσαν διάφορες ε, πτυχές του ελέγχου των προϊόντων αυτών καπνού. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα, ιδιαίτερα στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών, στον ε, χώρο που δραστηριοποιούμε εγώ για τον καπνό. Και η συνεργασία με τις ε, μονάδες του Όλαφ Διαφέρει ανάλογα με τη μονάδα, δεν μπορώ λοιπόν να γενικεύσω. Όμως μπορώ να πω ότι η πρόοδος είναι αργή αλλά σταθερή. Δυστυχώς πολύ αργή όμως. Και κατά την άποψή μου τα κράτη-μέλη είναι αυτά που βγαίνουν χαμένα και αυτός που κερδίζει είναι το οργανωμένο έγκλημα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι φραγμοί και τα προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Τώρα, τελευταία ερώτηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένους ε, παράγοντες. Υποθέτω ότι αναφέρεστε σε νομικές πτυχές. Όχι, λοιπόν, εμείς ε, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στα παράνομα εργοστάσια κατασκευής. Ελπίζω να έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας, όμως σας θα δεχτώ και άλλες ευχαρίστω. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιού. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Σε προηγούμενες ε, συζητήσεις, αυτήν εδώ την Επιτροπή, υπήρξαν κάποιοι που εξέφρασαν υποψίες για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον Όλαφ και την Ευρωπόλ. τις αρχές επιβολής νόμου των κρατών μελών και την καπνοβιομηχανία. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι ενδεχομένως αντιπαραγωγικό στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και ότι αυτή η έλλειψη καλής ανταλλαγής πληροφοριών εμποδίζει. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, νομίζετε πως είναι βάσιμες αυτές οι υποψίες. Να κρινίσω κάτι. Εννοείται τις πληροφορίες που μας δίνει η καπνοβιομηχανία που δίνει στον Όλαφ και την Ευρωπόλ. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. Αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν συναντήσεις με εκπρόσωπους των αρχών επιβολής ενόμου και της καπνοβιομηχανίας και συζητήθηκε μια κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Εσείς ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από αυτές ε, τις συναντήσεις, μπορούμε ως αποτέλεσμα να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Ακούσαμε και από τον κυρία Γκίλμορ ότι ενδεχομένως η καπνοβιομηχανία έχει συμφέροντα στο παράνομο εμπόριο. Εσείς ε, τι θεωρείτε πως ε, έχουν αποκομίσει οι εκπρόσωποι της καπνοβιομηχανίας από αυτό. Ναι, έχουμε ήδη καλέσει τους εκπροσώπους καπνοβιομηχανίας και σε ανοιχτές και σε κλειστές συνεδριάσεις και συναντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συμμετέχουν διότι ξέρουν απ' έξω το τι ακριβώς γίνεται, ποιες οδοί χρησιμοποιούνται και προσπαθούμε να πάρουμε όσες πληροφορίες ε, μπορούμε από αυτούς, να τις επαληθεύσουμε και να τις μεταβιβάσουμε και στις αρχές επιβολής νόμου των κρατών μελών. Σίγουρα είναι η καπνοβιομηχανία μια πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών και και εγώ ίδιος δεν θα είχα τόσο καλά αποτελέσματα στην, ε, στις μελέτες μου αν δεν χρησιμοποιήσω τις πληροφορίες που είχα. Δεν μπορώ να τις αγνοήσω, διότι δεν μπορώ να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ερευνές μου χωρίς αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκρέσλη έχει στήσει το λόγο μία ακόμη φορά. Μάλιστα και εμένα με απασχολεί αυτό το ζήτημα των δεδομένων. Τι ακριβώς δεδομένα είναι αυτά τα οποία λαμβάνετε. Είναι δεδομένα τα οποία εσείς μπορείτε να επαληθεύσετε, δεδομένα τα οποία εσείς ζητάτε από την, ε, το, τους καπνοπαραγωγούς και ποια είναι η νομική βάση την οποία χρησιμοποιείτε για να πάρετε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Όχι. Μπορείτε να απαντήσετε. Ή ο κύριος Φλόρεντς αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι. Κύριε Πιού, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε. Η Ευρωπόλη δεν έχει κάποια συμφωνία επίσημη, κάποια συνεννόηση με την καπνοβιομηχανία. Συναντιόμαστε συχνά και συζητούμε θέματα τα οποία μας ε, απασχολούν για να πάρουμε τις ε, αναγκαίες πληροφορίες, αντλούμε στοιχεία από διάφορους ε, παρόχους και όταν οι ίδιοι καπνοπαραγωγοί μας δίνουν τις πληροφορίες ζητούμε να μας το στείλουν και προσπαθούμε να επαληθεύσουμε τα στοιχεία αυτά, τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Φυσικά είναι περιορισμένες οι δυνατότητες ε, που έχουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό και πάρα πολλές περιπτώσεις εξάλλου είναι και εμπιστευτικές, είναι απόρριτες και είναι κάπως ε, μονόδρομος αυτή η ροή των ε, πληροφοριών. Έρχεται πρόστα εμάς, αλλά προσπαθούμε με τα δεδομένα που έχουμε να αποκομίσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα του τι γίνεται. Συλλέγουμε λοιπόν πληροφορίες, τις συνδυάζουμε από τις αρχές επιβολής νόμου, από το, εμπόριο και έχουμε μία βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλα αυτά και την οποία διαχειρίζεται ο Όλαφ. Αυτό λοιπόν το σύνολο μπορεί να μας δώσει και μια πολύ καλύτερη εικόνα και να μας βοηθήσει στο να προσανατολιστούμε σε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένους στόχους. Και αυτό μπορούμε μετά να το μεταφέρουμε και στα κράτη-μέλη. Ζητούμε λοιπόν εμείς αυτά τα δεδομένα. Συνδυάζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένοι κόμβοι, συγκεκριμένα σημεία, γιατί εμφανίζονται αυτά τα παράνομα προϊόντα στο α και όχι στο β μέρος και έτσι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε τις αρχές να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Η κυρία Γκρέσλε έχει και μια επιπλέον ερώτηση. Είναι πραγματικά συναρπαστικό αυτό. Είναι πολύ συναρπαστικό να δούμε ποιο είναι μέρο του προβλήματο και, ποια είναι, και ποιο είναι μέρο τη λύση. Μα είπατε ότι το 50% του λαθρεμπορίου γίνεται από την ίδια την καπνοβιομηχανία. Εάν λοιπόν το πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και η λύση, έχουμε σοβαρές δυσκολίες. Υπάρχει πρόβλημα. Εσείς μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το 25% του λαθρεμπορίου γίνεται όντως από την καπνόβιομηχανία και ε, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να εργαστούμε αξιόπιστα και να πάρουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Κάντενμπαχ, παρακαλώ. Ναι, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλε, να συμπληρώσω. Εάν το 25% των ε, λαθρέων προϊόντων προέρχεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόλοιπο ποσοστό. Το υπόλοιπο ποσοστό από πού προέρχεται και πώς ε, δημιουργείται από τους ε, επίσημους, από τους παραγωγούς, τους καπνοπαραγωγούς, από τους διαναμητές. Πώς μπορείτε εσείς να εντοπίσετε από πού προέρχεται. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Επίσης, υπάρχει Λέωνα, και περισσότερη η εντύπωση ότι οι μεγάλες εταιρείες παράγουν χαρτί, χαρτί τσιγαρόχαρτο το οποίο μπορεί και να διοχετευτεί για παράνομη κατασκευή τσιγάρων, για παράνομα τσιγάρα. Μπορείτε εσείς να μας το επιβεβαιώσετε. Μάλιστα. Ζήτησε το λόγο και ο ε, εκπρόσωπος της ε, GDI. Παρακαλώ. Όχι της Imperial, με συγχωρείτε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Adrian Welsh είναι το όνομά μου, εκπρόσωπος της Imperial. Να σας εκθέσω και την άποψη και την οπτική γωνία της δικής μου επιχειρήσης. Εμείς θεωρούμε πως είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Σας έδωσα πριν ένα παράδειγμα του τι δουλειά ακριβώς κάνουμε και σας ανέφερα και μια συγκεκριμένη ε, μάρκα τσιγάρων που παράγεται στην Ουκρανία. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν με πολλές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Όλαφ και με τα κράτη-μέλη. Και ένα παράδειγμα αυτών είναι ότι έχουμε κάποιες ε, επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου ε, παράγονται τέτοια παράνομα προϊόντα. Για παράδειγμα, συνεργαστήκαμε με το Βελγικό Τελωνίο και με τον Όλαφ για μια κατάσχεση, τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων τσιγάρων που είχε γίνει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έρχονταν από την Κίνα. Και οι πληροφορίες ήρθαν από το απεσταλμένο μας στο, ε, στην Κίνα. Ένα εμπορευματοκιβώτιο κατασχέθηκε στο λιμάνι της Μπρίζ, στην Μπρίζ, από το βελγικό τελωνίο και μετά ανακαλύψαμε ότι στο ίδιο σκάφος υπήρχε και ένα δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο με ελεύθερα τσιγάρα. Δεν είμαι φυσικά ειδικό στο πώ λειτουργεί... λειτουργούν οι αρχές της επιβολής νόμου. Όμως το ποσοστό που κατασχέθηκα ήταν 116 εκατομμύρια τσιγάρα καθώς και 16 εμπορευματοκιβώτια με παράνομα αρώματα αυτό πραγματικά ήταν ένα τεράστιο φορτίο και ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του πώς συνεργάζομαστε και πόσο καλά συνεργάζεται η καπνοβιομηχανία με τις αρχές επιβολής του νόμου. Υπάρχουν φυσικά πολλές ε, κατηγορίες ε, για εμάς, όμως υπάρχουν και πολλά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι συνεργαζόμαστε καλά. Και αυτό είναι ένα ακόμα ε, ένας ακόμα λόγος για τον, γιατί θέλουμε να θεωρούμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλόρεντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν σκιώδης εισηγητής της ε, κοινοβουλευτική μου ομάδας για την οδηγία για τον καπνό και πραγματικά με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι είστε μέρος της λύσης λέτε πως είστε μέρος της λύσης, από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Εύχομαι, λοιπόν, να είναι όντως έτσι τα πράγματα και να συμμετέχετε ενεργά στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πάνω από 20 χρόνια ασχολούμαι εδώ στο Κοινοβούλιο με αυτό το θέμα και ποτέ μέχρι τώρα, ποτέ άλλο το μέχρι τώρα δεν μου έχουν πει τόσα ψέματα για αυτό το πράγμα και πραγματικά ε, έχω παρατηρήσει ότι όσο ωραία και κομψά ρούχα να φοράνε και όσο ωραία λόγια και αν λένε τόσο πιο επικίνδυνοι είναι και τόσο πιο ε, πολύ, ε, τόσο περισσότερο ψεύδονται. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει οι συλλήψεις που έχουν γίνει στην Ιταλία, για παράδειγμα, σε όλη την επικράτεια της Ιταλίας, είναι, είναι κάτι απίστευτο. Το λαθρεμπόριο είναι καλπάζων και πραγματικά αυτό που βλέπω είναι ότι όσον αφορά την ίχνηλασιμότητα των ενεργειών των, του εμπορίου αυτού, έχω μάθει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει καλή συνεργασία. Για παράδειγμα, αυτά που έχω μάθει από τα γερμανικά τελωνία είναι ότι η συνεργασία είναι γενικά καλή και σε άλλες φορές... Ε, όχι, το... Εσείς τι έχετε να πείτε, ποια είναι η δική σας εμπειρία από τις τελωνιακές αρχές. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πιού, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, νομίζω η ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε στην αρχή είχε να κάνει με, το, ε, με την επαλήθευση των ε, στατιστικών στοιχείων. Η Ευρωπόλ δεν συλλέγει η ίδια στοιχεία για κατασχέσεις. Έχουμε ομάδα που κάνει ανάλυση των δεδομένων σχετικών με το οργανωμένο έγκλημα. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω πάνω σε αυτό, αλλά εμείς λαμβάνουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και όπως είδατε και από την παρουσίαση και το Project Star, λαμβάνουμε αυτά τα στοιχεία, τα εξετάζουμε, αλλά ακόμα και να διαφωνούμε με αυτά και να αμφιβάλλουμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη πηγή στοιχείων. Τώρα, επόμενη ερώτηση του κυρίου Κυρκεκάρτη ήταν για τα προϊόντα καπνού και τα εργοστάσια παραγωγή. Όταν φτιάχνει ένα παράνομο εργοστάσιο, λοιπόν, τα προϊόντα που χρησιμοποιεί είναι είτε εισαγόμενα. Είτε εισάγεις δηλαδή ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ε, παραγωγή τσιγάρων, είτε όχι, είτε είναι κάτι που υπόκειται σε ελέγχου, είτε κάτι παράνομο. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο σε περίπτωση που κάποια στατικά στοιχεία διακινούνται νόμιμα να ελεγχθούν. Και πολύ δύσκολο τομέα στον έλεγχο είναι ε, ο καπνός τα καπνά που είναι ακατέργαστα και διακινούνται για την παραγωγή τσιγάρων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να εντοπίσει τους παραγωγούς πώς διακινούν το προϊόν τους και για ποιους σκοπούς. Και νομίζω πως η άλλη ερώτηση είχε να κάνει με την συνεργασία με τα γερμανικά τελωνία. Κύριε Φλόρεντς. Με τη συνεργασία. Ναι. Ναι, επαναλαμβάνω ότι όταν επεξεργαζόμουν τα δεδομένα που είχα λάβει από τα γερμανικά τελωνία, είδα αυτή την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, θεωρούσαν τα τελωνία μη αποδεκτή και Θεωρούσαν λοιπόν πως αυτή η προσέγγιση δεν είναι σωστή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εσάς να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για την συνεργασία των γερμανικών τελωνίων με την υπηρεσία σας. Αν είναι καλή ή όχι. Έχουμε έναν σύνδεσμο των ε, τελωνίων στην Ευρωπόλ. Και μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας με ορισμένες περιοχές της Γερμανίας είναι καλύτερη από κάποιες άλλες. Δεν υπάρχει κάποια ενιαία προσέγγιση. Κάποιες περιοχές είναι καλύτερες στη συνεργασία, κάποιες όλες. Φυσικά και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και πιστεύω πως ένα από τα προβλήματα είναι ότι οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ακολουθήσουν πολλές διαφορετικές ε, προσεγγίσεις και αυτό είναι το πρόβλημα κυρίως δεν υπάρχει κάποια ενιαία προσέγγιση. Και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είχαμε παρατηρήσει το ίδιο πράγμα. Κάποιες, με κάποιες αρχές είχαμε καλύτερη συνεργασία, με κάποιες όχι. Επίσης, ε, οι ίδιες οι αρχές διαφέρουν. Μπορεί τα τελωνία να συνεργάζονται καλύτερα μαζί μας, αλλά οι αστυνομικέ αρχές όχι τόσο καλά. Μπορούμε, μπορώ όμω να σα πω ότι συνεργαζόμαστε καλά θα ήθελα να υπάρχει ακόμα καλύτερη συνεργασία, όχι μόνο με τις γερμανικές αρχές, αλλά και με τις αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών. Αλλά βλέπω ότι όλοι επιθυμούν μια καλύτερη συνεργασία. Και όταν συνεργαζόμαστε με κάποιο κράτος μέλος, δεν αναλαμβάνουμε εμείς ε, την ε, οργάνωση των επιχειρήσεων, αλλά συμμετέχουμε. Επίσης υπήρξε μια ερώτηση για, τους, ε, καπνο, για την καπνο, τους καπνοπαραγωγούς και αν υπάρχει κάποιο σχετικό μνημόνιο. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πράγμα. Πιστεύουμε πως η, η έλλειψη αυτού είναι κάτι καλό. Δεν, δεν λαμβάνουμε, δεν έχουμε κάποια έσοδα από αυτούς, δεν έχουμε κάποιες... Ε, τέτοιες σχέσεις, αλλά ελπίζουμε πως οι σχέσεις μας θα βελτιώνονται με την καλύτερη συνεργασία. Και πιστεύω πως η έλλειψη κάποιας τέτοιας συμφωνίας, κάποιου τέτοιου μνημονίου ε, διατηρεί αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πιού για την απάντησή σας σε όλες τις ερωτήσεις και πιστεύω πως κρατήσαμε το χρόνο διάγραμμα πάρα πολύ καλά. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στον τέταρτο ομιλητή, στον Λέσο Εκπαρτολιομιέτσικ από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας για το παράνομο επόριο καπνού στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ορίσατε. Και μπορείτε να αρχίσετε μόλις τελειώσουν και οι τεχνικές προετοιμασίες. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie i możliwość e, wypowiedzi w tak σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Καταρχήν θα σας μιλήσω για το παράνομο εμπόριο, το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού. Έχω συνεργαστεί με τον καθηγητή Τσιτσοβίτς και φυσικά εγώ θα περιοριστώ στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης τι καινούριο συμβαίνει στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέσα διαθέτουμε σήμερα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Όπως ξέρετε, το ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και το πιο μακρύ σύνορο, χερσαίο σύνορο και η χώρα μου είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τα σύνορα με την Πολωνία είναι ίσως και ο πιο σύντομος δρόμος για τα λαθρέα τσιγάρα που μπαίνουν από την Ανατολή στη Δυτική ε, Ευρώπη. Σκοπός αυτού του λαθρεμπορίου βεβαίως είναι να εισαχθούν παράνομα αυτά τα τσιγάρα. Θα πρέπει επίσης να δούμε και το ρόλο των ε, χώρων ε, διακίνησης αλλά και των χώρων από τις οποίες περνάνε όλα αυτά τα τσιγάρα. Η Πολωνία έχει αναπτύξει πάρα πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση αυτού του λαθρεμπορίου. Άκουσα αρκετές ερωτήσεις που κάνατε στους προηγούμενους ομιλητές που αφορούν τις πηγές των παράνομων τσιγάρων που βρίσκουμε στη δική μου χώρα. Πρέπει να σας πω ότι πολύ ισχυρή θέση κατέχει τα τελευταία χρόνια η ε, Λευκορωσία μεταξύ άλλων χωρών. Παλιότερα ο πρωταρχικός ρόλος παίζονταν από την Ουκρανία, κατόπιν τη Ρωσία, το Καλίνιγκρατ. Σήμερα όμως πρέπει να πούμε ότι πρωταρχικό ρόλο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων παίζει η τον Μπελαρού στη Λευκορωσία. Ο ρόλος των άλλων ανατολικών χωρών είναι περιθωριακός. Σε εμά στην Πολωνία περίπου το 60% των παράνομων τσιγάρων που εισάγονται προέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε από την Λευκορωσία. 60% και πολύ πρόσφατα χάρη στις έρευνες που διεκπαιρεώσαμε και στην αποτελεσματικότητα των διοκτικών αρχών της Πολωνίας στα σύνορα, διαπιστώσαμε ότι έχει μετακινηθεί το σημείο εισόδου προς δυσμάς της εισόδου παράνομων τσιγαρέτων στην Δυτική Ευρώπη, συγγνώμη, λίγο πιο νότια. Έχουμε ε, τον τελευταίο καιρό διεκπαιρεώσει πάρα πολύ επιτυχημένες ε, επιχειρήσεις τα τελωνία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διοκτικές αρχές έχουν καταφέρει να πλήξουν σημαντικά αυτό το λαθρεμπόριο. Έχουμε επίσης ιδιαίτερα ενισχύσει αυτή την δράση μας μετά το 2004. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι εγκληματίες προσαρμόζονται βεβαίως πάντα στην αποτελεσματική μας δράση. Γι' αυτό και όπως σας είπα έχει μετακινηθεί το σημείο εισόδου των ε, παράνομων τσιγάρων λίγο πιο νότια. Επίσης παρατηρούμε διαφορετική μορφή εισόδου, δηλαδή εισάγονται όλο και περισσότερα αποξηραμένα φύλλα καπνού, καθότι μετά το 2008 δεν μπορούν να ελεγχθούν με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι ε, αντικείμενα των ίδιων ρυθμίσεων. Φύλλα καπνού λοιπόν είναι το νέο παράνομο εμπόριο. Διαφορετικά κανάλια, διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικά προϊόντα. Βλέπουμε ότι ο έλεγχος στα σύνορα και η χρηματική στήριξη από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη ο εξοπλισμός των πολωνικών διοκτικών αρχών με νέο τεχνικό εξοπλισμό μας έχουν επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά έχει ε, βοηθήσει και τους ε, εμπόρους λαθρέων τσιγάρων να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους και να εξισορροπήσουν το κέρδος τους. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων πρέπει να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ενισχύσει μόνο μία συγκεκριμένη περιοχή, ένα συγκεκριμένο σύνορο, ενισχύοντας τους ελέγχους εκεί. Το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπως ξέρετε, δεν ε, γίνεται μόνο διασυνοριακά από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών. Εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπετε παράνομα τσιγάρα, τα οποία παράγονται στη χώρα μας, παράγονται στην Πολωνία και πολλούνται στην Πολωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εντοπίσουμε τη δράση μας όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ενισχύσουμε τους ελέγχους και στο εσωτερικό των χωρών Τι κάνουν ακριβώς οι διακινητές λαθρέων τσιγάρων. Για να μειώσουν το διαφυγόν τους κέρδος, αυξάνουν, πολλαπλασιάζουν τις αποστολές τσιγάρων, μειώνοντας τον αριθμό των τεμαχίων. Υπάρχουν ανώτατα όρια για τον έλεγχο εμπορευμάτων. Μειώνοντας λοιπόν τον αριθμό των τσιγάρων μιας αποστολής, μειώνονται και τα στατιστικά στοιχεία, αν θέλετε. Είναι κάτι που θεωρείται λιγότερο σημαντικό πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο ε, για την πάταξη των λαθρέων εμπορικών δραστηριοτήτων, αλλά και όσον αφορά τα έσοδα των κρατών. Χίλια φορτηγά γεμάτα με τσιγάρα είναι το διαφυγόν κέρδος. Τρία δισεκατομμύρια ζλότη για τη χώρα μας. Και ένα κόστος το οποίο βεβαίως αυξάνεται αν κάποιος συμπεριλάβει και τις θεραπείες όλων αυτών που έχουν ε, αρουστήσει εξαιτίας του τσιγάρου. Η καταπολέμηση λοιπόν αυτών των λαθρέων δραστηριοτήτων είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον γιατί βλέπουμε πόσο εύκολο είναι κάποιος ο οποίος εμπλέκεται σε μια παράνομη δραστηριότητα να έχει διακλαδώσεις και σε άλλα παράνομα εμπόρια. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων και πώς ε, οι έλεγχοι στα σύνορα έχουν αποτελεσματική δράση και στους ελέγχους τους ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών μας. Βλέπετε επίσης την ίδια δαφάνεια. Το λαθρεμπόριο, το παράνομο εμπόριο, αλλά και πολλές ε, άλλες δυνατότητες παραγωγής, εργοστάσια παραδείγματος χάρη, που ξεκινούν παράνομα, αλλά διοχετεύονται κατόπιν στο νόμιμο δίκτυο μιας χώρας. Οι παράνομες πρακτικές, όπως σας είπα και προηγουμένως, προσαρμόζονται, εξελίσσονται και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δύο πρωτόκολλα που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Πρόκειται για μία σύμβαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω και την οδηγία που αναφέρεται στα προϊόντα καπνού και που περιέχει κάποιες διατάξεις, κάποια στοιχεία για την παράνομη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Το σύστημα Track and Trace Επίσης, αποτελεί ένα τμήμα αυτού του οπλοστασίου καταπολέμησης της λαθρέας διακίνησης προϊόντων καπνού. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, όπως ακριβώς και το πρωτόκολλο για την εξάλληψη του λαθρεμπορίου καπνού. Πρόκειται για ένα από τα πρωτόκολλα που περιέχει τις πιο σημαντικές διατάξεις του αρθρο 8. Παραδείγματο χάρη γνωρίζετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου, το σύστημα track and trace προϊόντων καπνού. Θεωρώ λοιπόν ότι ο εντοπισμός όλων των προϊόντων καπνού, όλων των παράνομων προϊόντων καπνού, παραποιημένων προϊόντων καπνού, ο εντοπισμός των προϊόντων για εισαγωγή, για εξαγωγή και για τοπική κατανάλωση. Είναι απαραίτητο εδώ να υπάρχουν ειδικέ ενδείξεις για τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για την εξαγωγή για αυτών που θα πρέπει να παραμείνουν σε μια τοπική αγορά. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τους ελέγχους. Το πρωτόκολλο αυτό ορίζει με μεγάλη σαφήνεια ότι η παρακολούθηση και η έλεγχη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμπλέκουν τους εκπροσώπους της βιομηχανίας καπνού. Το πρωτόκολλο βεβαίως υπεγράφει από 30 χώρες και έχει τεθεί σε ισχύ. Υπάρχουν και άλλες πτυχές όσον αφορά την καταπολέμηση των λαθρέων τσιγάρων που συμπεριλαμβάνουν την ε, θέση σε ισχύ και την ε, εφαρμογή του track and trace. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τα κείμενα αυτά τον ε, Οκτώβριο του 2013. Η αναγραφή στα προϊόντα καπνού ενδείξεων που αφορούν την κατανάλωση των προϊόντων αυτών, καθώς και η ένδειξη όσον αφορά το έλεγχο, τον το, το ποιον ελέγχει και το κατά πόσο ελέγχονται οι διάφορες ε, τοπικές βιομηχανίες παραδείγματος χάρη είναι η παρακολούθηση της ε, αλυσίδας διάθεσης αλλά και κατασκευής. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ε, διαπραγματεύσεων των τριών τελευταίων μηνών, από τον Οκτώβριο δηλαδή μέχρι σήμερα, μπορέσαμε να επεξεργαστούμε τα κείμενα αυτά και να αφαιρέσουμε κάποια σημεία τα οποία ήταν ασαφή. Κατά την άποψή μου υπήρχαν ε, σημεία ασαφή τα οποία δίνουν δυνατότητες στους ε, παραβαίνοντες να παρεκκλίνουν των κειμένων ή να χρησιμοποιήσουν παραθυράκια, όπως παραδείγματος χάρη η πρόβλεψη συμμετοχής των εκπροσώπων της καπνοβιομηχανίας στην ε, διεργασία ελέγχων. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Ή παραδείγματο χάρη τις ενδείξεις χωρίς πιστοποίηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιος μπορεί να τυπώσει χαρτονομίσματα. Ότι η δυνατότητα εκτύπωση χαρτονομισμάτων μπορεί να δοθεί σε κάποιον χωρίς πιστοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι θέματα ασφάλειας. Σε καμία περίπτωση το κείμενο δεν θα πρέπει να δίνει τέτοιου είδους ε, δυνατότητες. Επίσης το θέμα των βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν υιοθετήσει τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές. Ε, γιατί, ε, παραδείγματος χάρη, μια χώρα μπόρεσε να είναι πιο αποτελεσματική. Ο εντοπισμός των προϊόντων, ο εντοπισμός από την παραγωγή μέχρι την πώληση. Επίσης βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική και η διενέργεια ελέγχων επί των ε, διαφόρων φορέων και οργανισμών, ποιος διεκπεραιώνει τους ελέγχους, ο εντοπισμός των προϊόντων από τη στιγμή που εμφανίζονται στην αγορά, γιατί εάν ε, περιμένουμε να διατεθούν Όπως ξέρετε υπάρχει το φαινόμενο του περάσματος ενός προϊόντος από την νόμιμη στην παράνομη αγορά ή και αντίστροφα. Ο ρόλος λοιπόν των ελέγχων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όλα αυτά τα στοιχεία αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της συχνηλασιμότητας αλλά και των ελέγχων και θα πρέπει πάντα, όπως σας είπα, να ξεκινούμε από την αρχή. Δηλαδή, να υπάρχει ένδειξη στα πακέτα τσιγάρων, όπως ακριβώς και σε άλλα έγγραφα ασφαλείας, επαναλαμβάνω όπως τα χαρτονομίσματα, με εμφανή ή κρυμμένα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν και στον καταναλωτή να αναγνωρίσει ε, το προϊόν, αλλά και στους ε, υπεύθυνους για τη διεκπαιρέωση των ελέγχων να διαπιστώνουν την χώρα προέλευσης, ε, το εργοστάσιο παραγωγής των τσιγάρων. Αυτά λοιπόν τα ενδεικτικά στοιχεία, οι μάρκες εμφανείς οι πιο κωδικοποιημένες θα πρέπει να είναι εύκολο να εντοπιστούν. Με, επαναλαμβάνω την υποχρέωση αυτό να γίνεται στην πηγή της κατασκευής και όχι όταν φτάσει ένα προϊόν στα σημεία πώλησης. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια αυτών των ενδείξεων. Να μπορεί κανείς να καταλάβει ποιος έχει παράγει και πότε έχει παραχθεί αυτό το τσιγάρο. Και αυτό βεβαίως ξεκινάει με μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, υπεύθυνου για τους φόρους κατανάλωσης, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα μπορούν να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν τα προϊόντα αυτά σε όλη την αλυσίδα διάθεσης και πώλησής τους στην αγορά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αν κάποιος ε, κλέψει παραδείγματος χάρη μια σφραγίδα ή ένα σύστημα ασφαλείας για τον, ε, την αναγραφή ενδείξεων πάνω στα πακέτα, αυτό θα πρέπει αμέσως να γίνεται αντικείμενο ενημέρωσης και να αλλάζει η αρμόδια αρχή αυτό το, αυτή τη σφραγίδα, παραδείγματος χάρη αυτή την ένδειξη, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραποίηση πακέτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχουν ειδικέ ενδείξεις στα πακέτα ή στις συσκευασίες ε, που περιέχουν παραπάνω από ένα πακέτο. Δεν είναι δυνατόν όταν γίνεται έλεγχος, παραδείγματος χάρη σε ένα κοντέινερ ή σε ένα φορτηγό, να ανοίγει ο ελεγκτής, ο τελωνιακός, το κάθε πακέτο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες με ένα τρόπο ο οποίος να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τεχνολογία, να ανοιχνεύσει εάν υπάρχουν ε, οι ε, ενδείξεις στα χαρτοκιβώτια ή στις συσκευασίες περισσότερων πακέτων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με ένα σκάνερ ή με κάποιον άλλο τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα στα τελωνία. Αυτό που θα πρέπει επίσης να μπορεί να ελέγχεται είναι ότι τα προϊόντα τα οποία ελέγχονται είναι αυτά που θα έπρεπε να βρίσκονται σε αυτό το κοντέινερ. Να μπορεί δηλαδή να ελεγχτεί η πραγματική ύπαρξη των προϊόντων που αναγράφονται. Όχι μόνο δηλαδή ότι πρόκειται για ένα γνήσιο τιμολόγιο, αλλά και ε, ότι το προϊόν το οποίο μεταφέρεται στο συγκεκριμένο κοντέινερ είναι το προϊόν το οποίο ε, έχει αρχικά προβλεφθεί. Τα συστήματα ελέγχου στα σύνορα αλλά και τα συστήματα ελέγχου στο εσωτερικό μιας χώρας θα πρέπει να γίνονται με ένα ομοιογενή τρόπο, με έναν εξοπλισμό ο οποίος θα πρέπει να επιτρέπει στο διανομέα να αποδείξει την αξιοπιστία του ή το κατά πόσο μεταφέρει γνήσια, νόμιμα ε, προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να πρόκειται για εξοπλισμό που να μπορεί να εντοπίσει την γνησιότητα των προϊόντων. Ο έλεγχος λοιπόν βασίζεται στη μάρκα των τσιγάρων και στις ενδείξεις οι οποίες πιστοποιούν τη γνησιότητα. Και βεβαίως, εάν πρόκειται για παραποιημένο προϊόν, να μπορεί πολύ εύκολα με ένα σκάν, με ένα κωδικό, να ε, επαληθεύσει κανείς ότι πρόκειται για γνήσια ή παραποιημένα προϊόντα. Επαναλαμβάνω πολλές φορές πρόκειται για γνήσια προϊόντα τα οποία όμως διακινούνται με παράνομο τρόπο για να μην υποβληθούν παραδείγματο χάρη στους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Ή ένα προϊόν το οποίο κανονικά έπρεπε να διατεθεί στην κυπριακή αγορά και το οποίο βρίσκεται σε μια άλλη αγορά. Το σύστημα track and trace κανονικά έχει και άλλες δυνατότητες και άλλα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανείχνευση και τον εντοπισμό των ε, παραποιημένων προϊόντων. Από τη στιγμή που κάποιος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα track and trace και αυτό θα εγκατασταθεί στις μονάδες παραγωγής, στα εργοστάσια παραγωγής, ο έλεγχος ε, θα ακολουθεί το προϊόν σε όλη την αλυσίδα διακίνησης παραγωγής και πώλησης. Εάν μια κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, αυξήσει του ειδικού φόρους κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ και αυξήσει την ίδια ώρα και τις δυνατότητες απάτης, με το σύστημα εχνηλασμότητας track and trace αποφεύγεται η ε, διαφυγή και η απάτη προς τις φορολογικές αρχές μετά το πρώτο έτος χρησιμοποίησης αυτού του συστήματος, πρέπει να σας πω ότι έχει διαπιστωθεί μια αύξηση των φορολογικών εσόδων που φτάνει μέχρι το 30%. Και αυτό όσον αφορά τα ε, τσιγάρα, τα πινοπνευματόδη, αλλά και τα προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας. Αυτό ασφάνει, αυξάνει συγγνώμη, και την ασφάλεια για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, αλλά και την αύξηση των εσόδων για τους κρατικούς ε, προϋπολογισμούς. Ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αυτό οφείλεται στην ε, χρησιμοποίηση του συστήματος Track and Trace και εδώ βλέπετε τρία παραδείγματα τριών κρατών που χρησιμοποιούν ήδη αυτό το σύστημα. Την Τουρκία και την πολιτεία της Καλιφόρνιας και βλέπετε στη διαφάνεια ότι τα έσοδα για τον κρατικό προπολογισμό αυξήθηκαν κατά 30% στις περιπτώσεις αυτής. Το λαθρεμπόριο μειώθηκε κατά επέκταση κατά 30%. Οκτώ παράνομα εργοστάσια τσιγάρων ε, έκλεισαν και αυτό χάρη στην ε, εφαρμογή αυτού του συστήματος. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζουν σε μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 50% την ε, ύπαρξη αυτών των ε, στοιχείων εντοπισμού στα πακέτα, ακόμα και αν αυτό αυξήσει την τιμή των τσιγάρων. Τελειώνοντας και συμπερασματικά θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν το πρωτόκαλο SCTC είναι ίσως και η σημαντικότερη δυνατότητα αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων μας. Θα πρέπει να αποτελέσει κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί και από μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης κυρίως προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που ανήκουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Αυτό θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τον τελεσματικότερο έλεγχο σε χώρε όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία. Η οδηγία που αφορά τα προϊόντα καπνού ελπίζω να συνεχίσει να βελτιώνεται και να μπορούμε να συμμορφωθούμε όσον αφορά τις διατάξεις αυτής της οδηγίας και το πρωτόκολλο για την πάταξη του παράνομου εμπορίου. Το θέμα της εχνηλασιμότητας, το σύστημα track and trace, πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σας εξήγησα, ελέγχουμε την παραγωγή, την διάθεση στο εμπόριο και αυξάνουμε και την ασφάλεια εντοπισμού αυτών των, των γνήσιων προϊόντων καπνού. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι βεβαίως και η διαφάνεια, η δημοσίευση των στοιχείων και των δεδομένων για το παράνομο εμπόριο αλλά και για το νόμιμο εμπόριο. Η κυρία Γκίλμορ αναφέρθηκε με πολλά στοιχεία ε, για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα εγώ να σας πω ότι όλες οι υπηρεσίες, τελεωνιακές και άλλες διοκτικές αρχές στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων όπως νέα σκάν. Το πρόγραμμα Ηρακλής ε, περιέχει τέτοιες δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρτολόμητη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Όσον αφορά το χρόνο που διαθέτουμε, έχουμε λίγο ξεπεράσει το χρόνο ομιλίας ε, για το θέμα σας, αλλά βεβαίως μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε όποιον θέλει να κάνει ερωτήσει. κυρία Γκρέσλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήμασταν στα σύνορα μεταξύ Καλίνγκραντ, στα σύνορα της Πολωνίας. Πήγαμε επίσης και στη Βουλγαρία, στα σύνορα Βουλγαρίας, Ελλάδας, Τουρκίας. Και είχαμε την εντύπωση ότι δεν είχαμε πάει στο σωστό σημείο για τα τσιγάρα, για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Μάλλον πρόσφυγες είδαμε εκεί παρά λαθρέα τσιγάρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνονται οι έλεγχοι, υπάρχουν άλλα σημεία εισόδου, άλλοι τρόποι διακίνησης που δεν Έχω και άλλες δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Είπατε ότι το θέμα των παραποιημένων φύλων καπνού είναι κάτι που μας απασχολεί. Πρόκειται εδώ για κάποιο κενό το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε όσον αφορά την νομοθεσία μας. Και έχω την εντύπωση ότι το θέμα του καπνού που πουλιέται ως καπνός και τα, παρα... και τα παραποιημένα τσιγάρα τα οποία ουσιαστικά κατασκευάζονται από τον ακατέργαστο καπνό και πώς αυτό μπορεί να καλυφθεί από νομικής απόψεως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακή αυτή η παρουσίαση και πολύ συγκεκριμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εννέα, αν δεν κάνω λάθος, στάσεις που μας κάνατε. Μία παρατήρηση και κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο ε, πρωτόκολλο SCTC ε, ε, πόσα κρατημέλη περιλαμβάνονται, ε, μήπως υπάρχει κενό, υπάρχει διαδικασία κύρωσης η οδηγία για το καπνό. Εδώ είναι πιο ευαίσθητο το θέμα για τα προϊόντα καπνού. Ε, το αρχικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν καλό. Όσον αφορά το track and tracing, ε, βάση κάποιων τροπολογιών που υπέβαλα με την κυρία Γκρέσλε, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε τα θέματα αυτά στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μετά υπήρχε η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο των Υπουργών, όπως μας είπατε, ε, αποδυναμώθηκε το κείμενο και φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Ε, μετά από τον τριμερή ε, διάλογο συνήφθη μια συμφωνία. Σήμερα στις 3 θα ψηφίσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κατόπιν το θέμα θα περάσει στην Ολομέλεια. Ελάχιστες κατά την άποψή μου είναι οι πιθανότητες να αλλάξει το κείμενο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο το μέλλον και να ε, πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει με αυτό το θέμα του track and trace. Είμαι πεπισμένος ε, ότι όσα μας είπατε είναι απόλυτα πιστικά, αλλά έχω τον εξή φόβο. Ε, στη μάχη με τους γίγαντες του καπνού υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι καταβάλουν ένα ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη Ε, βάση μιας κάποιας μορφής συμφωνίας και υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο τμήμα της συμφωνίας το οποίο αφορά τη διαδικασία του track and tracing. Ε, υπεγράφησαν ε, το 2004 ε, συμφωνίες με την PNR, με την Philip Morris και δύο χρόνια αργότερα μας είπανε πολύ ωραία πράγματα για το track and trace και τελικώς τα αποτελέσματα ε, στην Πολωνία είναι αυτά που μας παρουσιάσατε μόλις. Τι έγινε λοιπόν με αυτές τις συμφωνίες για τον καπνό. Εφαρμόστηκαν. Το track and trace εφαρμόστηκε. Ε, μήπως ε, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό το σύστημα από ό,τι περιμέναμε. Αυτή η ερώτησή μου. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κύριο Σεντεκάρτ. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Σε συνέχεια της ερώτησης της κυρίας Γκρέσλε, ναι, όντω εκ μέρου τη Επιτροπή υπήρξε μια επίσκεψη στο Καλίνιγκραντ και είδαμε ένα τελωνιακό σταθμό με μια πολύ σύγχρονη μονάδα ε, ελέγχου και έμοιαζε και με ένα μικρό χωριό. Μας έδειξαν επίσης και έναν ε, χώρο εργοστασιακών ε, προδιαγραφών ε, στην οποία γινόταν αποσυναρμολόγηση οχημάτων για να δούμε κατά πόσον υπήρχε λαθρέα διακίνηση προϊόντων. Ξέρουμε όλοι ότι όταν υπάρχει συνεργείο αυτοκινήτων υπάρχει πάντα διαρροή λαδιών και λοιπά, διαφόρων υγρών. Εκεί ήταν όλα πεντακάθαρα σαν να μην είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ ο χώρος για να γίνει από συναρμολόγηση οποιοδήποτε αυτοκινήτου. Yep. My name is Jakob Rasmussen from Copenhagen. Jakob Rasmussen από την Κοπενχάγη. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπαρτολο... Μπαρτομιέτσικ. Είχαμε μια μερίστη διάταξη πριν από τα Χριστούγεννα, όπου ε, αναφερόταν ότι ήσασταν ε, υπεύθυνο ε, επιχειρήσεων στη ΣΥΚΠΑ και σήμερα λέτε ότι είστε εκπρόσωπος κάποιου πανεπιστημίου. Και όλες οι διαφάνειες που είδαμε σήμερα, οι παραπομπές σε προϊόντα, οι παραπομπές σε τελωνία, είναι της εταιρεία σας. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία, αν συμφωνείτε. Ίσως αυτό να μην είναι το μόνο διαθέσιμο σύστημα για το track and trace και κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε και κάποιες ε, ανοιχτές ε, δυνατότητες, όπως για παράδειγμα το TS1, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για track and trace. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο ε, και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ανοιχτές πηγές προς όφελος των φορολογουμένων στην Ευρώπη, διότι το λαθρεμπόριο δεν είναι μόνο πρόβλημα που αφορά τον καπνό και την παραποίηση, αλλά πρόκειται και για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Ε, είναι ο πνευματόδη, ε, τρόφιμα και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να μας πείτε κατά πόσον εσείς είστε εκπρόσωπος κάποιου οργανισμού. Ε, είμαι εκπρόσωπος μιας ιδιωτικής επιχείρησης, της Factical Corporation. Factual Corporation. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Αν δείτε τη μελέτη την οποία δημοσίευσε το Τμήμα Πολιτικές, θα δείτε στο βιογραφικό του κυρίου Μπαλτομιατζίκ ότι εργάζεται και για μια ιδιωτική επιχείρηση. Υπάρχει ένα βιογραφικό σημείωμα για τον κύριο Μπαλτομιατζίκ. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της γενική Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. από αυτά που ακούσατε για τα θέματα και τις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ντόμινικ Νίκολς, ε, τμήματάρχης ε, του τμήματος 4 της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, που μεταξύ άλλων ασχολείται και με τον έλεγχο του καπνού. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό αυτό εργαστήριο είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον για πολλούς από εμά. Με τα χαράς να σας πω δύο λόγια για το άρθρο 14. Η κυρία Γκρέσλε νομίζω ότι μίλησε με τον Γενικό Διευθυντή μου εχθές και ήθελε να πούμε δύο λόγια για το άρθρο αυτό. Ελπίζουμε η αναθεωρημένη οδηγία για τα προϊόντα καπνού μαζί με το άρθρο 14 να ε, εγκριθεί τις επόμενες εβδομάδες. Οι συζητήσεις του τριμερούς διαλόγου όπως εξηγήθηκε ήδη ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο. Και αυτό το οποίο είναι προφανές για μας από πλευράς DigiSanco σήμερα είναι ότι το λαθρεμπόριο έχει πάρα πολλές όψεις. Και βεβαίως εσείς σήμερα νομίζω ότι ε, συζητάτε κυρίως το θέμα της φοροδιαφυγής ε, και από ε, το διαφυγόν κέρδος, οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά, τα οποία φυσικά είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικές πτυχές όλες αυτής της συζήτησης, αλλά εμείς από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ τα βλέπουμε και από ένα άλλο πρίσμα, το πρίσμα της δημόσιας υγείας. Το λαθρεμπόριο μας ενδιαφέρει κυρίως όσον αφορά το κατά πόσον ε, υποσκάπτει την ομοθεσία μας ε, για τα συστατικά και την ε, επισήμανση των προϊόντων και κατά πόσον η πρόσβαση σε προϊόντα καπνού είναι πιο εύκολη για το 70% των νέων ανθρώπων που καπνίζουν, διότι 70% των καπνιστών ξεκινούν κάτω από τα 18 τους και συνεχίζουν από εκεί και πέρα για όλη τους τη ζωή. Ε, δεν θα πρέπει βέβαια να σας εκπλήσει το γεγονός ότι εμείς ως DG Sankon θεωρούμε ότι η δημόσια υγεία είναι η πιο σημαντική. Περισσότερο μας ενδιαφέρουν οι 700.000 άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν καθημερινά ε, λόγω του τσιγάρου πρόωρα. Και θα ήθελα να το συνδυάζω αυτό με μια πάρα πολύ σημαντική διευκρίνηση. Ο βασικός στόχος της νέας οδηγίας δεν είναι η δημόσια υγεία, είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία διανέμονται στην ευρωπαϊκή αγορά συμμορφούνται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σχετίζεται λοιπόν κυρίως με τη νομική βάση της οδηγίας το θέμα αυτό. Η νέα οδηγία κάνει μια απόπειρα να αντιμετωπίσει όλα τα αίτια του λαθρεμπορίου, ε, λαθρεμπόριο, παραποιημένα, παράνομα λευκά και αυτό γίνεται με χρήση δύο μέσων του συστήματος Track and Trace και ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας ε, στις συσκευασίες. Σήμερα θα επικεντραθώ στο σύστημα track and trace, διότι προς τα εκεί οδεύουν και οι ερωτήσεις σας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τους ακρογωνιαίους λήθους οποιοδήποτε συστήματος προσπαθεί να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο, όπως δηλώνεται και στο πρωτόκολλο κατά του παράνομου εμπορίου, το οποίο ε, συνάφθη, ε, συνάφθη το 2012. Το σύστημα track and trace το οποίο διαθέτουμε βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Το άρθρο 14 θεμελιώνεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το σύστημα track and trace, ε, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά φυσικά θα πρέπει να αποκλείει το τελευταίο σημείο, το λιανεμπόριο, διότι δεν χρειάζεται να έχουμε στοιχεία από τους χιλιάδες ε, ή εκατομμύρια λιανεμπόρους που πολλούν τσιγάρα. Δεν χρειάζεται να γίνει επαλήθευση του συστήματος εκεί, διότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ. Δεν γίνεται εκεί άλλωστε η απάτη. Ε, εξετάζουμε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, διότι τα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε βεβαίως ε, λαθρέα τσιγάρα τα οποία προέρχονται από εξωτερικό, αλλά τα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται είναι ευρωπαϊκό εμπόριο και κυρίως ε, διαμεθοριακό εμπόριο. Ε, κάτι ακόμα, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα track and trace σε επίπεδο συσκευασία. Και αυτό γίνεται μέσω ενιαίου αριθμού αναγνώριση, ο οποίο ε, βρίσκεται επάνω στη συσκευασία. Και το πρωτόκολλο λέει ότι απαιτείται αυτό προκειμένου να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο. Ε, βεβαίως θα πρέπει από εκεί και πέρα να μπορούμε να έχουμε συνολικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε ε, να ζητούμε από τον οποιονδήποτε να σαρώνει απλώς ε, τα πακέτα. Θα πρέπει να γίνεται σάρωση ε, είτε σε παλέτες είτε σε μεγάλες συσκευασίες, σε εμπορευματοκιβώτια. Υπάρχει βέβαια αυτός ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης και πάνω στα πακέτα. Ε, ο δεύτερος πυλώνας του άρθρου 14 είναι ένα σύστημα εθνικού ελέγχου και αυτό ε, δεν θα πρέπει να έχει καμία επιρροή από την ίδια την καπνοβιομηχανία ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική επιρροή. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει με τη, να λειτουργήσει με τη συνδρομή όμως της καπνοβιομηχανίας. Το ε, πρωτόκολλο το λέει σαφώς, είναι ένα σύστημα κρατικού ελέγχου και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από τρίτη στον εξωτερικό παράγοντα, αλλά η ανεξαρτησία είναι εξίσου σημαντική και το άρθρο 14 λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία για παράδειγμα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ε, ε, μελλοντικής οποιοδήποτε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο συμβιβασμό, όπως σας είπα, επετέχθη μεταξύ των δύο συνομοθετών το Δεκέμβριο και πρόκειται για πολύ μεγάλο επίτευγμα. Εμείς φυσικά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτούμε τον συμβιβασμό και θα πρέπει να επισημάνω ότι οι συνομοθέτες ε, είχαν ε, ευθύ εξ αρχής παρόμοια άποψη όσον αφορά τους στόχους ε, και όσον αφορά και τις έννοιες και τα μέσα που θα χρησιμοποιούνται και νομίζω ότι οι δύο συνομοθέτες συμφωνούσαν επίσης ως προς τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 14 και ε, ως προς το γεγονός ότι αυτό είναι ο κρογωνιαίος λήθος, αλλά δεν θα αποφασιστούν τώρα οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν ε, μέσω εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατά εξουσιοδότηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί φυσικά να βοηθήσει ως συνήθως. Ε, ξεκινήσαμε με μια πολύ σημαντική μελέτη για τις τεχνικές δυνατότητες που μας παρέχονται για την δημιουργία ενός συστήματος track and trace από πέρσι και η μελέτη φυσικά θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2014 και επί τη βάση αυτής της μελέτης θα αποφασίσουμε. Δεν θα καθορίσουμε τώρα ότι υπάρχει μία και μόνη τεχνική λύση και θα πούμε ότι αυτή είναι η λύση της επιχείρησης Α ή της Β ή της Γ. Θέλουμε να κάνουμε μια διεξοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση και κατόπιν να αποφασίσουμε και μόνο τότε ε, να κρίνουμε ποια είναι η κατάλληλη λύση. Δεν υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο αποτέλεσμα ότι το σύστημα ΣΥΚΠΑ, για παράδειγμα, ε, προέχει ε, ή θα αγνοήσουμε το σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η ίδια η καπνοβιομηχανία. Υπάρχει ένα σύστημα της Φίλιπ Morris, για παράδειγμα. Θέλουμε να κάνουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και κατόπιν να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο και από τεχνική και από οικονομική σκοπιά. Θα λάβουμε όλα τα στοιχεία και κατόπιν θα αποφασίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Τώρα, τι μελιγενέστε. Καταρχάς, ε, θα προχωρήσει επίσημη έγκριση, ελπίζουμε ότι αυτή θα γίνει πολύ σύντομα. Η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει σήμερα και αναμένεται να ψηφιστεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια το ε, κείμενο, επομένως ε, σε ελάχιστες εβδομάδες σίγουρα πριν από τις ευρωεκλογές θα έχουμε ε, ένα τελικό εγκεκριμένο κείμενο και κατόπιν θα ε, υπάρξουν προτάσεις για τις εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις κατεξουσιοδότησης κατά πάσα πιθανότητα στη διάρκεια του επόμενου έτους. Νομίζω ότι με αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη παρουσίασή μου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μετά χαράς να σας απαντήσω. Αλλά να σας πω απλώς και μόνον ότι ε, συγχαίρω και τους δύο συνομοθέτες, διότι εργάστηκαν πάρα πολύ αποτελεσματικά στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Ήταν ίσως μία από τις πιο γρήγορες ε, συζητήσεις για ένα τόσο ακαθόδες από πολιτική σκοπιά ζήτημα και είμαστε ευγνώμονε για τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο για να επιτευχθεί τόσο σύντομα η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις, πολλές δηλώσει. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω απαντώντα στην πρώτη ερώτηση σχετικά με τον ακατέργαστο και τον αποξηραμένο καπνό και το πώς επηρεάζεται από αυτόν το παράνομο εμπόριο. Καταρχάς η απορρίθμιση το 2008 με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε την, τον την ανεξέλεγκτη παραγωγή καπνού και φύλων καπνού. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι στο νόμο αυτό, όμως κανένας δεν ελέγχει τους παραγωγούς και διανομής ακατέργας του καπνού. Τα κράτη-μέλη τα οποία είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τώρα ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα φύλλα καπνού. Αλλά και τα ακατέργαστα φύλλα καπνού αυτό που θέλουμε είναι ένα καλύτερος έλεγχος έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το φαινόμενο αυτό. Ωστόσο, έγκυται στη, στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και στο πώς αυτά θα αντιδράσουν. Τα φύλλα καπνού παράγονται στην Ευρώπη και μπορούν να αγοραστούν εκεί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηχανήματα τα οποία διευκολύνουν την συσκευασία του αποξηραμένου καπνού, την παρασκευή τσιγάρων τσιγάρα τα οποία μετά διοχετεύονται στην αγορά. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικό να δούμε τι αποτελεί έγκλημα και τι όχι. Στην παρανομία υπάρχει, στην Πολωνία, με συγχωρείτε, υπάρχει ε, αυτό που ονομάζουμε ενδιάμεσος ένας μεσάζων ο οποίος δεν πληρώνει αυτόν τον φόρο κατανάλωσης ακόμα και τον φόρο αυτό τον ε, αναλαμβάνει ο τελικός αγοραστής. Αυτό το, έχουμε, αυτό το έχουμε συμπεριλάβει σαν πρόταση για την ε, σύμβαση πλαίσιο FCTC. Μέχρι τώρα το πρωτόκολλο αυτό έχει υπογραφεί από 54 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μόλις αρχίσει η διαδικασία κύρωσης. Μία χώρα έχει ήδη πράξει αυτό στις 10 Ιανουαρίου και έχουμε τελειώσει με τη συλλογή υπογραφών. Έχουμε λοιπόν δύο εβδομάδες μέχρι να κυρωθεί η σύμβαση. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει και ελπίζουμε να τέθει σε ισχύ 90 μέρες αφότου επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για τον καπνό. Τα παραθυράκια που προέκυψαν από τις αλλαγές. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να έχουν το, ε, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες για αυτά λύσεις. Ακόμα λοιπόν και αν η οδηγία περιέχει κάποιες ε, πιο αδύναμες διατάξεις, ελπίζω να μπορέσουν τα κράτη-μέλη τα ίδια να προσθέσουν πιο αυστηρότερες διατάξεις. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα track and trace, καταρχάς, ε, να σας πω ότι στην ε, συμφωνία αυτό που υπάρχει δεν είναι ένα παρόμοιο σύστημα. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Η βιομηχανία χρησιμοποιεί κάποια από αυτά τα συστήματα. Στην Ευρώπη Καμία χώρα δεν χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα track and trace και αυτό που αναφέραμε πιο πριν είναι κάποια, ε, κάποιες συστάσεις. Συστάσεις από άλλα κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βραζιλία για παράδειγμα, την οποία ανέφερα, Τουρκία. Αυτά είναι κράτη τα οποία έχουν παρόμοια συστήματα με το track and trace, τα ε, οποία το χρησιμοποιούν κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιθέτως έχει σταματήσει, έχει παγώσει αυτό το σύστημα λόγω των ε, πολλών υπογραφών που χρειάζονται. Δεν μπορούμε λοιπόν ακόμα να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σύστημα μέχρι ότου συμφωνήσουν όλοι. Τώρα, αν υπάρχουν προβλήματα εδώ, η έλεγχη των μεμονωμένων πακέτων τσιγάρων που έχει αναφέρει η καπνοβιομηχανία δεν είναι πάντα δυνατόν να γίνουν. Διαπιστώνεται η αυθεντικότητα του πακέτου, βέβαια με, αυτές, με αυτά τα συστήματα μπορούμε να δούμε τον ε, αριθμό, τον κωδικό του κάθε πακέτου και μετά να βρούμε στο ίντερνετ σε τι αντιστοιχεί. Και αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί μπορούν όντως να ελεγχθούν. Αυτά ως προς το σύστημα. Φυσικά ένα τέτοιο σύστημα δεν εφαρμόζεται, σας είπα ακόμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω όμως αυτό να γίνει σύντομα. Τώρα, η επόμενη ερώτησή σας είχε να κάνει με το τι γίνεται στα σύνορα, με τι έχουμε παρατηρήσει εμείς στα σύνορα. αναφέρατε το Καλίνιγκρατ και τους ελέγχους που γίνονται σε αυτοκίνητα που σταματούν. Στο Καλίνιγκρατ είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πριν από κάποια χρόνια. Τα τσιγάρα παρασκευάζονταν εκεί, όμως τώρα δεν έχουμε πια πρόβλημα ελαφραίων τσιγάρων από το Καλίνιγκρατ. Τώρα προέρχονται από αλλού, από τα, ε, από τα ανατολικά και χρησιμοποιούνται τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ως ένα τρίγωνο εισαγωγής λαθρέων τσιγάρων και το σύστημα αυτό αλλάζει κάθε λίγα χρόνια. Κάθε δύο-τρία χρόνια τα τσιγάρα αλλάζουν μέρος από το οποίο μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά είναι πολύ πιο συμφέρον οικονομικά να αλλάζει αυτό και να μετακινούνται αυτές οι δύο πιο προσταθητικά. Τώρα, ε, για την επόμενη ερώτησή σας. Συνήθως δεν απαντώ σε προσωπικές ερωτήσεις, όμως επειδή είμαστε ενώπιον μιας τόσο καλής ομάδα θα ήθελα να σας απαντήσω ότι η παρουσίαση αυτή έγινε μαζί με τον κύριο Ζόβιτς, τον καθηγητή του Ζόβιτς, Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό να παρουσιάσω την ε, μελέτη αυτή εκ μέρους μια ιδιωτική εταιρεία. Όχι, η έρευνα αυτή έχει γίνει μαζί με τον ε, καθηγητή ε, του Ζόβιτς και αυτό και έχετε εδώ. Τώρα, εάν, υπάρχει, εάν αυτό το σύστημα track and trace είναι το μοναδικό, νομίζω πως η απάντηση είναι προφανής. Δεν είχα στην μελέτη μου κάποια αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Αναφερόμουν μόνο στις βέλτιστες πρακτικές. Εάν ρωτάτε αν το σύστημα που δημιούργησε η δική μου εταιρεία είναι το μοναδικό, θα σας απαντήσω ότι είναι το μοναδικό σύστημα που χρησιμοποιείται από αρκετές χώρες για να γίνεται αυτός ο έλεγχος track and trace των προϊόντων καπνού. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπάρτολο Μιέτσεκ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις περιεκτικές και σύντομες απαντήσεις σας. Προτείνω λοιπόν τώρα για λόγους οικονομίας χρόνου να ζητήσουμε από το πέμπτο πάνελ να λάβει το λόγο. Έχουμε τρεις ομιλητές, τον Λουκ στην Χάνα και, στο, και τον Μίχαλ στο Κλώσα. Σας ζητώ λοιπόν να κάνετε την παρουσίασή σας. Έχουμε σχεδόν ετοιμάσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και μπορείτε να αρχίσετε. Καλημέρα σας. Έχουμε 15 λεπτά λοιπόν και θα σας παρουσιάσουμε μια έκθεση η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με τους δύο συναδέλφους μου, την Χαναρό και τον Μίχαλη Στοκλόζα. Ε, εργάζονται για την ε, Αμερικανική Αντικαρκυνική Εταιρεία, αλλά προέρχονται από την Τσεχία και από την Πολωνία ένα από τα προβλήματα του να είσαι τελευταίος ομιλητής είναι ότι πολλά από τα θέματα που θέλει να θίξει έχουν ήδη αναφερθεί από τους προηγούμενους. Έτσι λοιπόν, θα προσπαθήσω μαζί με τους συναδέλφους μου να σας παρουσιάσω συνοπτικά τρία θέματα. Μας ζητήθηκε να φτιάξουμε μια έκθεση για την αξιολόγηση της ε, στρατηγικής και του σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση ε, του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, να ε, εξετάσουμε την αναθεωρημένη οδηγία για τα προϊόντα καπνού και τις συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη και τέσσερις ε, μεγάλες καπνοβιομηχανίες. Πρώτο θέμα λοιπόν θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία της έκθεσης και κάποια θέματα ήδη αναφέρθηκαν κατά ε, την παρουσίαση της Άννα Γκίλμορ. Μας ζητήθηκε λοιπόν να εξετάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου και το πρώτο που παρατηρήσαμε ήταν ε, η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων. Υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα στη διάθεσή μας στην παρούσα πολιτική και βασιζόμαστε κυρίω σε δύο ε, δεδομένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τι εκατασχέσεις και στοιχεία που μα δίνει για τα πακέτα για τις συσκευασίες η Φίλιπ Μόρι. Είναι ίσω ενδιαφέρον να αναφέρω την προέλευση των προϊόντων αυτών καπνού. Κάθε φορά που κατάσχεται κάποιο τέτοιο προϊόν πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται και το ίδιο συμβαίνει και με τις έρευνες που κάνουν οι εταιρείε για τα άδεια πακέτα. Και Ούτε μάλλον το ένα ούτε το άλλο δεν επαρκούν για να κάνουμε μια σωστή εκτίμηση του παράνομου εμπορίου και της έκτασής του. Τώρα, όσον αφορά τα δεδομένα από το Project Star, να σας πω ότι στο project αυτό, στην πρώτη κιόλα σελίδα της ε, έκθεσης, αναφέρεται ότι η KPMG επιθυμεί να γνωρίζουν όλοι ότι η έρευνα που έγινε είχε σκοπό να... Ε, είχε γίνει κατόπιν εντολή τη Φίλιπ Μόρι και ζητήθηκε για να ανταπεξέλθει σε ειδικέ ε, απαιτήσει που γνωρίζει μόνο η Φίλιπ Μόρι, σε απόρριτα δεδομένα δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένα σημείο αναφορά και αυτό είναι η Φίλιπ Μόρι. Αναφέρεται λοιπόν ότι η έρευνα αυτή ζητήθηκε από την Φίλιπ Μόρις, από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα 27 κράτη-μέλη. Αυτό είναι λάθος και η πληροφορία αυτή πρέπει να διορθωθεί. Η δουλειά έγινε μόνο κατόπιν αιτήματος της Φίλιπ Μόρις και φυσικά κάποιες χώρες είχαν μεγάλα ποσοστά λαθρεμπορίου, όμως δεν συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι αυτό αυτή η έρευνα, αυτή η μελέτη δεν ε, μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικό δεδομένο. Είναι κάτι που έγινε για λόγους τους οποίους ε, μόνο η Φίλιπ Μόρις γνωρίζει και είναι εμπιστευτική. Υπάρχει ε, λοιπόν μια σύγκρουση συμφερόντων. Και η Όλαφ, ο Όλαφ μάλλον και η Ευρωπόλ δεν συμμετείχαν σε αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε εάν ε, συμφωνούν ή διαφοδούν με τη μεθοδολογία που ακολούθησε η ομάδα που έκανε τη μελέτη ή αν η μεθοδολογία αυτή ε, συμφωνεί με αυτά που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Η Άννα Γκίλ Μωρίδη σας έκανα μια εκτενέστατη παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι τα δεδομένα που στηλέχθηκαν ε, ήταν από πακέτα τσιγάρων. 10.000 ε, πακέτα σε, μεγαλ, σε μεγαλύτερες χώρες, 5.000 πακέτα σε μικρότερες ε, χώρες. Πολλοί εντυπωσιάζονται από αυτούς τους αριθμούς. Δεν είναι όμως αλήθεια. Εξαρτάται από το πού μαζεύει κανείς τα πακέτα. Αν για παράδειγμα τα συλλέξουμε εδώ στις Βρυξέλλες, γύρω από το, από το σταθμό Μιντή ή από κάποιο γήπεδο ποδοσφαίρου, θα βρει κανείς ένα μεγάλο αριθμό παράνομων πακέτων. Αν πάτε σε άλλες περιοχές θα βρείτε σχεδόν ε, τίποτα, θα βρείτε μόνο νόμιμα πακέτα. Πρέπει λοιπόν να δοθούν αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες και αφόσον η Public Star δεν τι δίνει δεν είναι αξιόπιστες. Το έγγραφο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν αναφέρεται στην Public Star, είναι δεδομένα που προέρχονται από τη βιομηχανία και να σας ε, πω ότι αυτό που αναφέρεται σε γενικές γραμμές είναι ότι το παράνομο εμπόριο αυξάνεται και ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση όταν εισαχθεί η νέα νομοθεσία για την, ε, για την ε, απλή συσκευασία. Χρησιμοποιούνται λοιπόν αυτά τα δεδομένα από τις κατασχέσεις για, και έχουν εκτιμηθεί απώλειες περίπου 10 δισεκατομμυρίων. Όμως δεν γίνεται να δοθούν αξιόπιστα δεδομένα για το παράνομο εμπόριο, διότι εξαρτάται η αξιοπιστία από πολλά δεδομένα, από τις ε, αρχές επιβολής του νόμου και τα δεδομένα, από τα δεδομένα που δίνονται από την βιομηχανία, από τις ε, κατασχέσεις που γίνονται και τον αριθμό των ε, τσιγαρών που κατάσχονται. Ας δούμε πρώτα τις κατασχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να δούμε και τι μπορούμε να μάθουμε από τον συνολικό παγκόσμιο ρυθμό κατασχέσεων των ε, τσιγάρων. το 2000 παρατηρήθηκαν οι περισσότερες κατασχέσεις και το 2000 ήταν η χρονιά ε, κατά την οποία η καπνοβιομηχανία είχε κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τότε και αργότερα 10 κράτη-μέλη ε, έκαναν μήνυση στην, ε, στις εταιρείες αυτές. Μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα τι έγινε στην Ιταλία. Στην Ιταλία το 1999 κατασχέθηκαν 2 δισεκατομμύρια τσιγάρα. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά πολύ σε, μέσα σε δύο χρόνια. Και προτού υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία. Και επίσης παρατηρείται μείωση των κατασχεμένων τσιγάρων ακόμα και τώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι κατασχέσεις μειώνονται, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες του Project Star οι κατασχέσεις αυξάνονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιόπιστα δεδομένα. να ασχολιάσω τώρα την πολιτική της Επιτροπής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε με, ε, με το πρωτόκολλο FCTC και την ε, εφαρμογή του. Ήμουν παρόν σε όλες τις σχετικές συναντήσεις από το 1998 ως εκπρόσωπος της ε, κυβέρνησης του Βελγίου και ως προσωρινός σύμβουλος του ΠΟΕ, ως μέλος μη κυβερνητικών οργανώσεων για το πρωτόκολλο λοιπόν FCTC μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχω παρατηρήσει πολύ στενά την ε, δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είχαμε κάποιο πρωτόκολλο μέχρι τώρα και να σας πω ότι όλα αυτά οφείλονται σε ένα πρόσωπο, οφείλονται στον ε, πρόεδρο τη Επιτροπή, ο οποίο κατέβαλε ο ίδιο τεράστια δουλειά για να καταφέρουμε να έχουμε στα χέρια μα αυτό, όχι μόνο διαπραγματευτικό έργο, αλλά και προωθούσε και ενημέρωνε για το πρωτόκολλο αυτό από το 2001. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ένα χρόνο με τα περιγράφει το πρωτόκολλο το 2012. 12 χώρες το έχουν υπογράψει μέχρι τώρα και μόνο μία το έχει επικυρώσει και πέρυσι ήδη πιστεύαμε ότι ο αριθμός αυτός θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Δεν συνέβη όμως αυτό. Όσον αφορά τη σύμβαση πλαίσιο τώρα, η, η συνθήκη που υπεγράφει το 2003 συμπεριλάμβανε 60 χώρες που το είχαν ε, υπογράψει και 23 που είχαν επικυρώσει το πρωτόκολλο και αυτές που δεν το επικύρωσαν ε, το έπραξαν αυτό γιατί δεν είχαν την ε, τεχνική δυνατότητα, δεν είχαν την εμπειρογνωμοσύνη και δεν είχαν και πόρους Και να σας πω για την έλλειψη πόρων ότι για το 2014 και 2015 τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας είναι γύρω στα 200.000 ευρώ, ένα πολύ μικρό ποσό δηλαδή. Επομένως, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και πλήρη ε, εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Τώρα οι δηλώσει που και τα στοιχεία που έχουμε από τον Όλαφ, από την Ευρωπόλη, από τις αρχές εφαρμογής του νόμου δείχνουν ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης παρασκευής. Τι χρειάζεται λοιπόν για να παρασκευάσεις παράνομα τσιγάρα γενικότερα. Θέλεις καπνό, θέλεις χαρτιά, χαρτάκια και θέλεις φιλτράκια. Ανέφεραν ήδη προηγούμενοι ομιλητές στον ακατέργαστο καπνό. Είναι ένα φορολόγητο ε, προϊόν το οποίο μάλιστα επιχορηγείται. Χρειάζεται λοιπόν ο έλεγχος του ακατέργαστου καπνού, διότι διαφορετικά, εάν ε, υπάρχει παντελής έλλειψη ελέγχου, θα συνεχιστεί το παράνομο εμπόριο. Δεν υπάρχουν λοιπόν προς το παρόν ε, μέτρα για να ελέγχεται ο ακατέργαστος καπνός, παρομοίως και με τα χαρτάκια και τα φίλτρα. Κάτι άλλο σχετικό με την πολιτική του Όλαφ είναι οι σχέσεις του Όλαφ με, τους, ε, με, τα γραφεία επαφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένας ε, απεσταλμένος στην ε, Κίνα από το 2011 μέχρι το 2012. Δεν ανεώθηκε όμως η σύμβασή του. Έχουμε επίσης και έναν εκπρόσωπο στην Ουκρανία. Έναν, μόνο έναν. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα όμως έχει 28 υπαλλήλου απεσταλμένους σε διάφορα σημεία του κόσμου. Και το έργο του Ηνωμένου Βασιλείου και η οργάνωση αυτή κατάφερε να αποτρέψει απώλειες ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους 28 διαφορετικούς ε, απεσταλμένους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της με έναν, ο οποίος δεν βρίσκεται και πλέον στην ε, Κίνα. Η Κίνα έχει δείξει προθυμία να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να λείπει από εκεί κάποιος ε, σύνδεσμος. Έπειτα, ε, όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, καταλαβαίνω γιατί η καπνοβιομηχανία ήδη από, τη, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 όταν εφαρμοστηκε η πρώτη οδηγία για τον καπνό εξέφρασε τις αντιδράσεις της και προειδοποίησε για την αύξηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων και προϊόντων καπνού. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την οδηγία για τον καπνό το 2001 αναφέρθηκε ότι εάν υπάρχει έλεγχος για την εξαγωγή τσιγάρων και αν υπάρχει περιορισμός στο περιεχόμενο πίσας και νικοτίνης και ε, μονοξιδίου του άνθρακα, αυτό θα οδηγήσει σε μαζικό λαθρεμπόριο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί, διότι έχουν, έχει μειωθεί και ο αριθμός των κατασχέσεων και αυτό φαίνεται. Όμως η Imperial Tobacco έχει κάνει μαζικές εξαγωγές προϊόντων τα οποία ήταν μόνο γνωστά ε, στην ε, Βρετανία σε χώρες όπως ε, οι χώρες της Βαλτικής Ανδόρα και το Λιχτενστάιν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για, τις, για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν εξαγωγές οι εταιρείες αυτές, αλλά πολύ λίγα δεδομένα που σχετίζονται με, την οδηγία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προϊό... πολλές έρευνες, όπως αναφέρθηκε, οι οποίες έχουν ζητηθεί από τις ε, ίδιες τις ε, καπνοβιομηχανίες. Ο μεγαλύτερος φόβος της καπνοβιομηχανίας είναι η απλή συσκευασία των τσιγάρων. Το πρόβλημα όμως ε, αυτό έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Το άλλο πρόβλημα είναι για τα τσιγάρα μενθόλης που εκρεμεί. Το πρόβλημα για τα τσιγάρα slim έχει επιληθεί. Τώρα, με τα τσιγάρα της μενθόλης τι θα μπορούσε να συμβεί. Ότι μπορούν οι καπνιστές αυτών των τσιγάρων να προχωρήσουν σε άλλες μάρκες ή να ε, ψάξουν αυτά τα τσιγάρα στη, στην παράνομη αγορά. Η περίοδος σταδιακής ε, κατάργησης των τσιγάρων αυτών έχει μειωθεί από τα 8 στα 6 χρόνια και αυτό που αναμένεται είναι οι καπνιστές των τσιγάρων μενθόλης να προσαρμοστούν και να αλλάξουν σε απλά, σε κανονικά τσιγάρα. Αυτό τώρα που πιστεύουμε εμείς είναι ότι οι χώρες οι οποίες έχουν πολύ μικρή κατανάλωση τσιγάρων μενθόλης δεν θα επηρεαστούν καθόλου από αυτήν την ε, απαγόρευση. Ε, ενδεχομένως υπάρξουν κάποιες ε, Επιτόσεις ε, και αλλαγέ σε χώρε που έχουν μεγάλη κατανάλωση τσιγάρων μενθόλης όπως η Πολωνία και η Φιλανδία. Έχουμε παρατηρήσει όμως ότι όσοι καπνίζουν τσιγάρα μενθόλης πολύ δύσκολα θα καταφύγουν σε λαθρέα τσιγάρα, σε παράνομα τσιγάρα. Ο, και ο τυπικός καπνιστής αυτών των τσιγάρων είναι γυναίκα, νέα, ενώ στην στη Φιλανδία αυτό, ενώ στην Πολωνία ο αντίστοιχος καπνιστής είναι άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας που ζει στην Ήπεθρο. Δεν αναμένουμε λοιπόν μια μεταστροφή του αριθμού αυτού των καπνιστών ε, τσιγάρων μενθόλη στην παράνομη αγορά. Στη χειρότερη περίπτωση το μόνο που θα συμβεί θα είναι μια απώλεια εισοδήματος για την καπνοβιομηχανία. Τώρα, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες που έχουμε με την ε, καπνοβιομηχανία, τα τελευταία 10 με 20 χρόνια διατηρώ στενές ε, επαφές με τον Όλαφ, και παρατήρησα ότι η μήνυση, η αγωγή αυτή που είχε κατατεθεί προ τι μεγάλε αυτές εταιρείε, τη Philip Morris για παράδειγμα, είχε μεγάλες επιπτώσεις στη μετέπειτα οργάνωση του παράνομου εμπορίου. Το 2004 και το 2007 οι αγωγές αυτές αποσύρθηκαν κατά της Philip Morris και της Japan Tobacco. Εδώ βλέπετε τον ε, Μίσελ Πετίτ που ήταν ο Γενικός ε, Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μετά έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Φίλιπ Μόρις. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρξε έτσι μία σύγκρουση συμφερόντων. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών λοιπόν των συμφωνιών του 2004 και του 2007 είχαμε δύο συμφωνίες συνεργασίας με την BAT και την Imperial το 2010. Κατέβαλαν λοιπόν κάποια χρηματικά ποσά στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μια συμφωνία για τα τσιγάρα τα οποία κατάσχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικά τους τσιγάρα. Εάν λοιπόν τα τσιγάρα αυτά κατάσχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνουν κάποιο ποσό ανάλογα με την ποσότητα που κατάσχεται. Τι βρήκαμε τώρα στις έρευνές μας για τα τσιγάρα Classic. Και επί τη ευκαιρία να πω ότι χαίρομαι πολύ που έχουμε και τον εκπρόσωπο της ε, εταιρεία εδώ. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να συλλέξουμε αρκετέ πληροφορίε για, για το πόσα τσιγάρα έχουν κατασκευθεί στην Ευρώπη. Είχα ακούσει μια παρουσίαση του Ιαν Βόλτον στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό το 2009, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρθηκε στο ποια τσιγάρα κατάσχονται περισσότερο στην Ευρώπη. Στην πρώτη θέση ήταν τα Μάλμπορο, στην τρίτη θέση ήταν τα Κλάσικ. Τα Classic είναι μία μάρκα της Imperial Tobacco. Το 2010, όπως είπα, υπήρξε συμφωνία με την Imperial, η οποία θα πλήρωνε με βάση τις κατασχέσεις τσιγάρων της εταιρείας της. Όμως το 2009, 10, 11 και 12 δεν ε, καταφέραμε να συλλέξουμε κάποια δεδομένα για τις κατασχέσεις στην, σε ορισμένες χώρες, στην Πολωνία. Τα κλάσικα όμως ήταν τα τσιγάρα τα οποία κατασχέθηκαν περισσότερο στη χώρα αυτή. Μόλις ε, πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας η έκθεση της Monitors από το 2013. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα Classic ήταν η δεύτερη, η δεύτερη δημοφιλέστερη μάρκα τσιγάρων για το 2012. Επίσης, σύμφωνα με τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Πολωνίας, όπου υπάρχουν παρόμοια στοιχεία. Ο εκπρόσωπο ε, λοιπόν τη Imperial μας ανέφερε ότι έχει σταματήσει η παραγωγή της μάρκας αυτής, της Classic, Και πραγματικά μετά από αυτά τα δύο στοιχεία που έχουμε πρέπει πραγματικά να μάθουμε τι συμβαίνει με τα classic. Δεν έχουμε λοιπόν αξιόπιστα στοιχεία και το πρόβλημα αυτό θα επιληθεί μόνο εάν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τις κατασχέσεις των τσιγάρων αυτών. Τα classic παραμένουν πρόβλημα. Τώρα, εάν η Imperial χρησιμοποιεί ένα άλλο εργοστάσιο κάπου αλλού για την παρασκευή τους, είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Εξακολουθούν όμως να πολλούν τα τσιγάρα αυτά, παρότι έχουν αποσυρθεί, Τα τσιγάρα όμως αυτά πολλούνται σε ορισμένα. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, δεν μπορούν λοιπόν να ε, θεωρηθούν ως παράνομα λευκά. Τώρα, όσον αφορά τις ε, πληρωμές ε, που προκύπτουν από τις κατασχέσεις. Πρέπει να δούμε ποιε εταιρείε είναι αυτές που έχουν καταβάλει πληρωμές. Δυστυχώ δεν έχουμε δεδομένα. Και πρέπει και ζητήσαμε και από τις 27 ε, χώρες το 2012 να μας δώσουν δεδομένα σχετικά με αυτά, λάβαμε όμως ε, απάντηση μόνο από 8 από αυτές. Ο κύριος Στάς ήδη ανέφερε ότι το πρόβλημα με την έκθεση Project Star, την οποία ζήτησε και πλήρωσε η Φίλιπ Μόρις, είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση αυτή το 92% των κατασκευμένων τσιγάρων είναι ε, απομιμής, είναι παραποιημένα. Όμως υπάρχουν δεδομένα που ε, λένε το ακριβώς ε, αντίθετο. Υπάρχει λοιπόν μια... Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Οι εταιρείε αυτές ε, δεν χρειάζεται να πληρώσουν αυτό... αυτά τα ποσά εάν αποδειχθεί ότι τα τσιγάρα είναι παραποιημένα. Και οι εταιρείε είναι αυτές που που θεωρού που που χαρακτηρίζουν τα τσιγάρα από μιμήσεις ή γνήσια. Έτσι λοιπόν, τα χαρακτηρίζουν ως παραποιημένα και ως απομιμήσεις για να μην χρειαστεί να καταβάλουν πληρωμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν Αντίθετε πληροφορίες. Η μία λέει 16% παραποιημένα, η άλλη 92% παραποιημένα. Οι μόνες πληροφορίες λοιπόν που έχουμε, που μπορούμε να θεωρήσουμε κάπως αξιόπιστες, είναι αυτές που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Και εδώ βλέπουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασχέθηκαν 460 εκατομμύρια τσιγάρα το 2012. Ένα μόνο εκατομμύριο από αυτά ε, μπορούσε να θεωρήθηκε γνήσιο, χαρακτηρίστηκε γνήσιο, οπότε κατέβαλαν και πληρωμές. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίστηκαν ως ε, παραποιημένα και έτσι οι εταιρείε δεν χρειάστηκε να καταβάλουν πληρωμές κατάσχεσης. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η βιομηχανία δεν, είναι, δεν έχει ευθύνη για αυτό το λαθρεμπόριο. Όπως σας είπα λοιπόν, λάβαμε απαντήσεις και πληροφορίες από 8 χώρες σχετικά με τις πληρωμές εκατασχέσεων. Η Εστονία, η Πολωνία και η Σλοβακία χρησιμοποιούν τα, τις αυτέ αυτές τα ποσά για να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ενώ τα, ε, οι ε, στο Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι άμεσες πληρωμές στον, στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που επίσης παρατηρήσαμε στην περίπτωση της Πολωνίας είναι ότι η βιομηχανία χρησιμοποιεί τα ποσά αυτά για διαφήμιση Αυτά λοιπόν ήταν εν ολίγης τα ευρήματα της έκθεσής μας. Είναι διαθέσιμη σε όλους και μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ. Θα προεδρεύσω για λίγα λεπτά, γιατί ο πρόεδρος αναγκάστηκε να βγει. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μία ερώτηση όσον αφορά την εξάλληψη, την κατάρριση του μηχανισμού. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και τους τρεις για την συνεισφορά σας. και για την προετοιμασία αυτής της παρουσίασης. Μιλήσατε για το πρωτόκολλο FCTC καταρχήν και σε μία από τις συστάσεις που μας παρουσιάσατε λέτε ότι θα πρέπει η διάδοση του καπνού, του τσιγαρόχαρτου, των φίλτρων θα πρέπει να ελέγχεται, θα πρέπει να περιοριστεί. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί σας, γιατί όταν μιλούσαμε για τις απάτες το 1997 ήδη, ήδη είχαμε μιλήσει για την ενίσχυση του ελέγχου και στα φίλτρα και για τα πακέτα και για τον καπνό αλλά και για τα έτοιμα τσιγάρα. Είχαμε μάλιστα πει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα είδος ειδικέ μηχανές, πιστοποιημένες μηχανές για την ε, κατασκευή των τσιγάρων, παραγωγή τσιγάρων. Αλλιώς μπορεί κανείς πολύ εύκολα να αρχίσει και να παράγει τσιγάρα σε παράνομα εργοστάσια. Ο κύριος Γιώσεν αναφέρθηκε επίσης στις κατασχέσεις και μας λέει, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν από αυτόν, ότι ουσιαστικά οι καπνόβιομηχανίες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα σαν γνήσια ή παραποιημένα. Και, και βεβαίως τίθεται το θέμα της ανεξαρτησίας. Μιλήσαμε προηγουμένως για το Scottish Institute που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Ηρακλής και ότι όταν μπει κανείς στην ιστοσελίδα αυτού του σκοτσέζικου οργανισμού δεν αναφέρεται τίποτα απολύτως που αφορά το τσιγάρο, το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δίθεν ανεξάρτητη έλεγχη οι οποίοι δεν πραγματοποιούνται εμένα μου δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα και όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτουμε. Άλλοι λένε 16% παραποιημένα τσιγάρα, άλλοι πάρα από 90%. Βλέπουμε ο Επίτροπος σε μέτα, ο οποίος στην ανακοίνωσή του μιλάει για τις συμφωνίες με την βιομηχανία καπνού και αναφέρεται ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν υπογράψει την συμφωνία και το κατά πόσο υπάρχει σημαντική μείωση αυτών που υπέγραψαν, των εταιριών που υπέγραψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία και αντίθετα, αυτοί που δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία γνωρίζουν μια αύξηση της τάξης του 58%. Αυτό το 58% που ανακοινώνει ο Επίτροπος στην δήλωσή του, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ε, ε, δικαιολογείται. Θα απαντήσω καταρχήν στην πρώτη ερώτηση που έχει σχέση με την Κίνα, της κυρίας Κρέσελ. Βασιζόμενοι στα στοιχεία του Βρετανικού Κοινοβουλίου το 2008 επισήμως σταμάτησε αυτή η δραστηριότητα από μέρους της Κίνας και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλα αυτά συνεχίζει να λέει ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες παράνομων προϊόντων, εμπορευμάτων έρχονται ακόμα από την Κίνα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Υπάρχουν ε, πάνω από τέσσερις ή έξι, αν θέλετε, υπεύθυνοι για τους ελέγχους για αυτό το συγκεκριμένο τόπο προέλευσης παράνομων εμπορίων. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο ε, κόστος. Η ερώτησή σας για τον ακατέργαστο καπνό και τα άλλα προϊόντα καθώς και για το πρωτόκολλο στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Εμείς ε, καταρχήν πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε κατά, αν κοιτάξει κανείς τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα διαπιστώσει και όταν διαβάσει την έκθεση του Όλαφ ή της Europol διαπιστώνει ότι υπάρχει παράνομη παραγωγή στην Ευρώπη, στο εσωτερικό της Ευρώπης, από προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί παράνομα και χωρίς να υποστούν κανένα ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι είμαστε κατά και να μην παραδεχόμαστε ότι υπάρχει τέτοια παράνομη παραγωγή στην Ευρώπη. Η απάντηση της Επιτροπής, αν ναι ή όχι, είναι αποτελεσματικές οι συμφωνίες. Στο έγγραφο της Επιτροπής, στη σελίδα 6, διαβάζουμε ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι ναι, είναι αποτελεσματικές οι συμφωνίες, διότι οι κατασχέσεις των άλλων εταιριών, των άλλων πολυεθνικών καπνοβιομηχανιών, οι τέσσερις και οι άλλοι, δηλαδή, συγκρίνουν τις κατασχέσεις και λένε ότι οι κατασχέσεις των άλλων εταιριών αυξάνονται κατά 58%. Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι έτσι κι αλλιώς όταν διαβάζω μια τέτοια δήλωση, γιατί όλοι ξέρουν ότι οι μεγάλες πολυεθνικές σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχουν μειωθεί Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά, βλέπετε τα στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς εδώ στην Ευρώπη, όπως και οι άλλες μεγάλες ήπειροι, γνωρίζουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα ξέρουμε ότι η παράνομη δραστηριότητα αυξάνεται και όλοι ξέρουμε ότι οι κατασχέσεις, τα στοιχεία για τις κατασχέσεις τα έχουμε από πολύ συγκεκριμένες πηγές. Όταν κοιτάξει λοιπόν κανείς τις ερωτήσεις, τις κοινοβουλευτικές, ποια είναι η μάρκα που, για την οποία έχουμε τις περισσότερες κατασχέσεις, η απάντηση είναι δεν έχουμε στοιχεία. Ενώ εδώ λένε ότι 58% είναι από άλλες εταιρείες. Άρα στοιχεία υπάρχουν, έχουν στοιχεία για την κάθε μάρκα ξεχωριστά, για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά και απλώς δεν θέλουν να μας τις δώσουν. Το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν τα στοιχεία για την κάθε εταιρεία, απλώς δεν θέλουν να μας τα δώσουν, ιδιαίτερα όταν αφορά τις κατασχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η ευρωπαϊκή πολιτική είναι αποτελεσματική ή όχι, γιατί δεν ξέρουμε σε τι στοιχεία βασίζεται. Uh, possibly to Προς αυτούς που είναι παρόντες από την Επιτροπή κάνω την ερώτηση. Πού βασίζεται αυτό το 58%? Επίσης το ίδιο θα ήθελα να ρωτήσω και για το Ινστιτούτο από την Σκοτία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Όσταν Ρον. Είμαι σύμβουλες στην Όλαφ ο κύριος Γιούσεν μίλησε για αυτό το 16% και για το 58%. Θα ελέγξουμε αυτούς τους αριθμούς και θα επανέλθουμε. Μπορώ επίσης να συζητήσω και διμερός μαζί του αν το επιθυμεί. Η δική σας ερώτηση για το θέμα των κατασχέσεων. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η σύμβαση αυτή που επεγράφει από τρία χρόνια με το Ινστιτούτο στη Σκοτία έγινε γιατί ήταν σε θέση να αναπτύξουν ένα σύστημα που μας επέτρεπε να βρούμε την προέλευση των προϊόντων καπνού. Δεν είμαι ειδικό για θέματα φύλων καπνού κτλ. αλλά μπορώ να σας πω ότι όταν κατεργαστεί αυτός ο καπνός, η περιεκτικότητά του σε χημικά και διάφορα άλλα στοιχεία φυσικά και αυξάνεται. Αυτές οι ουσίες, χημικές και άλλες, μπορούν να μας οδηγήσουν στην προέλευση του καπνού. Από άποψη δηλαδή πληροφοριών, ήταν πολύ καλή ιδέα να αποτανθεί κανείς σε αυτό το Ινστιτούτο το σκοτσέζικο με την έννοια ότι μπορούσαμε να εντοπίσουμε τα προϊόντα παραποίησης ε, ανάλογα με την σύνθεσή τους, τις χημικές ουσίες που περιείχαν και την προέλευσή τους, την Κίνα παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα στον ιστότοπό τους. Γιατί θέλαμε, και δεν το είπαμε εξάλλου καν στις πολυεθνικές εταιρείες αυτό, να θελήσαμε να διατηρήσουμε κατά κάποιο τρόπο διακριτικά αυτήν την επαφή με αυτό το Ινστιτούτο. Θελήσαμε να γίνει όσο πιο διακριτικά και ανεπίσημα γίνεται. Και Από τη στιγμή που υπάρχει κατάσχεση, ξέρετε ότι υπάρχει και η καταβολή ενός ποσού από μέρους των ε, εταιριών. Γι' αυτό και παίζει καθοριστικό ρόλο εδώ αν θα χαρακτηριστούν τα προϊόντα σαν γνήσια ή παραποιημένα, διότι το ποσό καταβάλλεται μόνο όταν πρόκειται για γνήσια προϊόντα. Και εδώ παίζει ιδιαίτερο ρόλο αν παραδείγματο χάρη ένα προϊόν είναι γνήσιο, αλλά χαρακτηριστεί παραποιημένο. Σε αυτή την περίπτωση εμεί ζητούμε να αποτανθεί κανεί σε εμά στον Όλαφ, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την έρευνα και να δούμε αν πραγματικά είναι παραποιημένα η γνήσια προϊόντα και για ποιο λόγο χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα, εάν ο σκοπός είναι ε, να αποφύγει μία επιχείρηση την καταβολή ενός ε, ποσού. Πρόκειται λοιπόν για μια διαμάχη που πολλές φορές μπορούμε να την διαλευκάνουμε. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα προϊόν το οποίο έχει κατασχεθεί, έχει χαρακτηριστεί σαν παραποιημένο. Εμείς κάνουμε την ανάλυση και βγαίνει χαρακτηρίζεται σαν γνήσιο. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να πάει σε ένα ανεξάρτητο εργαστήριο και να συμφωνήσει η επιχείρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρμόδια αρχή ότι θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση για να αποδειχθεί η γνησιότητα ημί των προϊόντων. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο σε επιστοποιημένους και κοινά αποδεκτούς οργανισμούς. Αυτή την περίπτωση είναι το Βρετανικό Δημόσιο Εργαστήριο Ανάλυσης. Και πραγματικά αυτό είναι η ευκαιρία για να διαλευκανθούν κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Εμείς ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας στείλουν ένα δείγμα από το κατασχεθέν προϊόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δεκπεριάσουμε περαιτέρω ελέγχους και να αποδειχθεί αν ναι ή όχι εδώ οι επιχειρήσεις παίζουν ε, ξεκάθαρο ρόλο ή όχι. Πρόεδρος, είμαστε ακόμα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Μία ερώτηση. Γιατί αυξήθηκε το όριο για τη Φίλιπ Μόρις. Ποτέ δεν είχαν πετύχει το προηγούμενο νοτατόριο. Και αν εδώ συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιου είδους ε, χειρισμοί όσον αφορά τα στοιχεία, γιατί το κάνατε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, λέει ο πρόεδρος. Μία ερώτηση. Μάλιστα έχετε το λόγο. Πολύ σύντομη ερώτηση. Τι λύσεις προτείνετε. Όσον αφορά την ανείχνευση και την ε, δίωξη, την πάταξη. Τι, τι λύσεις προτείνετε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να απαντήσει. Έχουμε το πρωτόκολλο για το λαθρεμπόριο και αν όπως ελπίζω συμβεί αυτό που θα συμβεί σήμερα το απόγευμα, το Κοινοβούλιο δηλαδή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υπερψηφίσει την ε, οδηγία, θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα όταν θα εγκριθεί η οδηγία για τη ε, προϊόντα καπνού. Αυτό θα σημαίνει ότι το 2019 θα υπάρχει πλέον ένα σύστημα το οποίο θα επιβάλλεται από την νομοθεσία, θα ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έχει φυσικά συνέπειες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιο σύστημα επισημώ. Θέλω να υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο ελέγχονται τα στοιχεία από τις αρχές και αυτό θα μπορεί να γίνει με την έγκριση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και θα υπάρχουν συνέπειες και για την υπογραφή και κύρωση πολλών άλλων ε, χωρών. Το πώς θα λειτουργήσει αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, βρισκόμαστε στην αρχή του 2014, σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις, αλλά ελπίζω ε, να έχουμε και κάποια πράγματα για το πρωτόκολλο για το παράνομο εμπόριο. Εκτός μικροφώνου η ερώτηση του ομιλητή. Δημοσίευσα ένα άρθρο δεν είναι σαφής η θέση μου για το ε, ε, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχεται και θα το διαχειρίζονται οι αρχές. Και για να είμαι σαφής, δεν θέλουμε, εγώ μάλλον δεν θέλω, ένα σύστημα Ε, όπως το Project Star για τα στοιχεία για το λαθρεμπόριο, το οποίο το ελέγχει η Φίλιπ Μόρις και το διαχειρίζεται η Φίλιπ Μέρις και στρεβλώνει και τα στοιχεία όπως επιθυμεί η Φίλιπ Μόρις αν κάτι ε, το διαχειρίζεται η καπνοβιομηχανία και υπάρχει ο ίδιος ο, σύστη, ο, ο έλεγχος της καπνοβιομηχανίας ε, για το σύστημα track and ε, trace, τότε είμαστε όλοι χαμένοι. Χρειαζόμαστε ένα ανεξάρτητο σύστημα και πρέπει να ελέγξουμε ποιο θα λειτουργήσει καλύτερα. Σας παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει διάλογος ούτε συνεντεύξεις εδώ στην αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εργαστήριο εδώ. Μπορείτε κάλλιστα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε εκτός αιθούσης. Εδώ στο εργαστήριο θέλουμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τελειώνει και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, ίσως θα μπορούσατε απλώς και μόνο να μας πείτε ποιος είστε. Ζητώ συγγνώμη, Άντωνη Μπολτάνοβιτς. Ε, εκπροσωπώ την ε, Matomat.po, μια στα σελίδα. Υπήρχε μια ερώτηση και προς τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σίγουρα. Έγινε αναφορά στην baseline θα πρέπει λίγο να ανατρέξουμε και στο πότε διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρις. Η διαπραγμάτευση έγινε από το 2001 μέχρι το 2004. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολες οι διαπραγματεύσεις όπως θα φαντάζεστε. Ήταν η πρώτη τέτοια συμφωνία και καταλήξαμε σε ένα αρχικό ποσό 90 εκατομμυρίων. Βέβαια θα πρέπει να ε, θυμόμαστε και το εξή. Όταν ε, δημιουργήθηκε αυτή η συμφωνία, είχαμε 15 κράτη-μέλη, μετά εντάχθηκαν 10 νέα κράτη-μέλη και το πρόβλημα ήταν ότι το ποσοστό λαθρεμπορίου και παράνομο εμπορίου στη χώρα αυτή ήταν πολύ ψηλό. Ε, κάποιες χώρες ε, αντιστοιχούν στο 40% της αγοράς. Στο μεταξύ συνάθησαν και άλλες συμφωνίες και είχαμε βασιστεί για το βασικό ποσό βάσει του μεριδίου αγορά και ε, είχαμε διαπραγματευτεί ένα ποσό των 50 εκατομμυρίων. ο κύκλο εργασιών τη Philip Morris είναι τριπλάσιο από τη BAT. επομένω. γι' αυτό είχαμε 90 εκατομμύρια για τη μία και 50 εκατομμύρια για την άλλη. Ποτέ βέβαια δεν φτάσαμε αυτό το ποσό των 90 εκατομμυρίων, ούτε καν το πλησιάσαμε, αλλά αυτό το οποίο θέλαμε ε, είναι να τα ανακλάτε γιατί ε, είναι 50 τα εκατομμύρια της BAT. Η Φίλιπ Μόρις έχει τριπλάσιο κύκλο εργασιών, γι' αυτό και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ποσά. Ε, ένα σχόλιο και για το Project Star, διότι ακούστηκαν πάρα πολλές επικρίσεις για το Project Star, ότι το χρησιμοποιεί η Φίλιπ Μόρις για να χειραγωγεί την κατάσταση και το καθεξής. Η Όλαφ σε καμία περίπτωση δεν έχει χρησιμοποιήσει το Project Star ως βάση για να καθορίσει ε, το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα 10 δισεκατομμύρια. Ε, το ποσό αυτό βασίζεται στις κατασχέσεις, μπορεί να μην είναι απόλυτα ορθά τα στοιχεία για να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα, αλλά αυτό χρησιμοποιούμε. Δεν βασιστήκαμε ποτέ στο Project Star. Το Project Star προέκυψε προκειμένου να καθορίσουμε αν τα νέα 10 κράτη-μέλη όταν εντάχθηκαν θα είχαν δικαίωμα να λαμβάνουν ε, πληρωμές για αυτές τις κατασχέσεις. Διότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο παράνομο εμπόριο στις χώρες αυτές και η Φίλιπ Μόρις ε, θεώρησε ότι ίσως ε, θα χρηματοδοτούσε και την έλλειψη ελέγχων σε ένα κράτος μέλος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησαμε το Project Star για να καθορίσουμε και συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη και συμφωνήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την KPMG για όλη τη μεθοδολογία. Το όλο σκεπτικό ήταν να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα εργαλείο, ένα εργαλείο για να καθορίσουμε αν τα κράτη-μέλη θα είχαν δικαίωμα σε πληρωμές για τις κατασχέσεις. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι θα ήταν με στοιχείο που θα μας έδινε πληροφορίες, που θα έδινε πληροφορίες στην Όλαφη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποτέ δεν θεωρήθηκε ότι το έγγραφο αυτό θα διατίθεται δημοσίως στο κοινό υπήρξε έτοιμα για πρόσβαση στα έγγραφα από κάποια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έλαβε τα έγγραφα και δεν τους αρέσει το περιεχόμενο. Δεν φταίμε εμείς όμως γι' αυτό η Φίλιπ Μόρις ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας είπε ότι δεν θα το δημοσιεύσει σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς διέρευσε, αλλά εμείς δεν το χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως όλη αυτή η ιστορία έχει ολοκληρωθεί, γιατί όλα τα κράτη-μέρη λαμβάνουν πληρωμές για τις κατασχέσεις και επομένως δεν εφαρμόζεται πλέον το μέσο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό λοιπόν φτάσαμε σχεδόν στο τέλος, σχεδόν στο στόχο μας. Να ευχαριστήσω όλους θερμότατα όσους συμμετείχαν εδώ. Και θα τώρα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ίνια Κρέσλα για τα τελευταία σχόλια. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ όλους. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε ε, τον ρόλο, το ρόλο ε, ε, το δικό σας ε, στη συμφωνία για τον καπνό και το μέλλον αυτής. Ε, μπορώ να πω ότι δεν είμαι και κατενθουσιασμένη με όλα αυτά που είδαμε, όμως ε, βλέπω επίσης ότι και η συμφωνία για τη διαφάνεια δεν έχει οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω πως αυτό έρχεται και μεταξύ άλλων επειδή όλα δεν έχει ασχοληθεί τόσο ενεργά με αυτό. Όμως πιστεύω πως ε, πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο τέλος. Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό χωρίς πρώτα να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για λεπτομέρειες, να συζητήσουμε για ποσά, για τα ποσά κατασχέσεων. Τα ποσά κατασχέσεων είναι αστεία στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε μιλάμε για ε, τριψήφιους ε, αριθμούς για, για δισεκατομμύρια δολάρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτό ε, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αναδιάρθρωση του Όλαφ και να δούμε το τι θα γίνει με την μονάδα για τα τσιγάρα. Η κατάργηση μιας τέτοια μονάδας θα έχει πάρα πολύ αρνητικέ συνέπειε, Ήδη είδαμε τι έγινε στην Κίνα με τον έναν υπάλληλο ο οποίος ε, μάλιστα αποχώρησε. Χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται από κοινού στρατηγική για να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο. Καταρχάς πρέπει πρώτα να ε, δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε το, το λαθρεμπόριο. Διαφορετικά μπορούμε να ξεχάσουμε τα, ε, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Έχουμε ένα κοινό συμφέρον, ένα κοινό στόχο και αυτός ο κοινό στόχος είναι η καταπολέμηση του ε, λαθρεμπορίου. Γι' αυτό χρειάζεται να συζητήσουμε, χρειάζεται να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού έχουν πάει όλα τα κονδύλια και τι γίνεται με, τα, με τις πληρωμές από τις κατασχέσεις. Πιστεύω πως θα ήταν καλό να λάβουμε επιτελούς μια οριστική ε, θέση και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αποφασιστικοί, να δράσουμε με αποφασιστικότητα έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε κάποια λύση στο τέλος του τούνελ. Είναι κοινό μας συμφέρον, όπως είπα, να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο και είναι επίσης ε, απαραίτητο γι' αυτό να συμμετέχουν όλοι και να συμμερίζονται όλοι τον ίδιο στόχο. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρέσλε. Τελευταίος έχει το λόγο ο εισηγητή. Να πω και εγώ δύο λόγια ε, δεν έχω και πολλά να πω. Ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ συναρπαστικές παρουσιάσεις. Ε, μας δώσατε και πολύ υλικό, ε, πολλά στοιχεία, ε, αριθμητικά στοιχεία και νομίζω ότι σήμερα το πρωί ακούστηκαν ε, πολλά πράγματα για τις προκλήσεις, για το τι πρέπει να γίνει. Όλα αυτά θα συγκεντρωθούν φυσικά σε ένα έγγραφο. Ε, δεν μπορούν να γίνουν πολλά όσον αφορά την νομοθεσία μέχρι το τέλος της ε, ε, φαντάζομαι ότι το επόμενο κοινοβούλιο ε, η επόμενη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα έχει πολλή δουλειά μπροστά τη. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα θέματα αυτά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο εργασία και θα έχουμε και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορεί λοιπόν να θέσει ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού στον αρμόδιο επίτροπο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα αυτά και θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ο νέος Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα καταπολέμησης της απάτης. Ε, πέρασε η ώρα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Ευχα... Αυτά από μένα. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Σε όλους όσους συμμετείχαν ευχαριστήσω και τον εισηγητή αλλά και τις τελωνιακές αρχές του Βελγίου που μας επέτρεψαν να σας φέρουμε εδώ στη μέση της αίθουσας αυτά τα προϊόντα κατασχέσεων γιατί θέλαμε να έχουμε και ένα απτό παράδειγμα αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο, όλους όσους ε, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Ίσως δεν αφήσαμε όλους τους εκπροσώπους των διαφόρων λόμπι να πάρουν το λόγο. Εμείς θέλουμε πραγματικά να επεξεργαστούμε όλες τις πτυχές γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό στην Ευρώπη.